διότι τότε τις διαβάζουμε εμείς στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή, για να δει αν είναι εφικτές οι ιδέες αυτές, αν έχουν, αν διαθέτουν νομική βάση. Έτσι έχουμε ένα πρώτο, μια πρώτη ας πούμε ιδέα για το εάν όντω θα μπορέσουν να λειτουργήσουν αυτές ε, οι ιδέες, αυτές οι προπαρασκευαστικές ε, δράσεις κ.ο.κ. Αυτά λοιπόν χρειάζεται να διαβαστούν στην Κομισιόν πριν από τις 29 Πέμπτου είδα ότι η Επιτροπή σας δραστηριοποιείται σημαντικά σε ό,τι αφορά τη χρήση της δυνατότητας και πιλωτικών ε, έργων και προπαρασκευαστικών δράσεων. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και εγώ, κύριε Γένσεν. Η Ιούτα Χάουκ. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, συμφωνώ με κάθε λέξη που ακούσατε από τα χείλη της Αν Γένσεν. Η Κομισιόν ασφαλώς δεν μπορεί να εργαστεί στην βάση των αριθμών που έφτιαξε στις 8 Δευτέρου το Συμβούλιο. Αυτό είναι σαφές. Ούτε μπορεί να βασιστεί στην πρόταση της Κομισιόν, ούτε άλλωστε μπορεί να βασιστεί στην δική μας πρόταση της ΣΟΥΡΕ που θα ήταν το καλύτερο για μας. Ενδεχομένως η Κομισιόν να πρέπει να κάνει τα όσα πρέπει να κάνει εφόσον δεν διαθέτουμε πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, άρα δηλαδή δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου, θα πρέπει τότε η Κομισιόν να εργαστεί στη βάση των οροφών του προπολογισμού του 2013... και να συνεχίσει το, με τον τρόπο αυτό. Νομίζω θα τα καταφέρει μέχρι τα μέσα Μαΐου. Τώρα, πιο συγκεκριμένα για την Επιτροπή Περιβάλλοντος και για τα όσα μας απασχολούν πιο ε, ειδικά, βρισκόμαστε μάλλον στον τελευταίο χρόνο του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου και των δύο προγραμμάτων, δηλαδή του προγράμματος ε, δράσεων για την υγεία και του προγράμματος περιβάλλοντος LIFE. Και θέλουμε βέβαια στο τέλος του έτους να διαθέτουμε προϋπολογισμό, ο οποίος να μας επιτρέπει να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και του χρόνου τις ε, πληρωμές για τις οποίες έχουμε δεσμευτεί ήδη. Άρα τα διάφορα προγράμματα τα οποία έχουν, για τα οποία έχουν αναλυφθεί, ανα, αναλυφθεί να μπορέσουν όντως να εφαρμοστούν. Αυτό ισχύει και για το LIFE και για το πρόγραμμα δράσεων στον τομέα της υγείας. Είμαι πεπισμένη ότι και φέτος θα αναλυφθούν ακόμη περισσότερες υποχρώσεις και επομένως χρειαζόμαστε τα αντίστοιχα κονδύλια. Τώρα, πιλωτικά προγράμματα και προπαρασκευαστικές δράσεις. Ευτυχώς εδώ οι συνάδελφοί μας έχουν λάβει την ενδιάμεση έκθεση της Κομισιόν το έγγραφο εργασίας που έχει συντάξει η Αν Γένσεν με τον φετινό εισηγητή το μόνο που μπορώ να πω εδώ είναι εξετάστε το προσεκτικά και ας στοχεύσουμε στα πιλωτικά προγράμματα τα οποία έχουν ήδη ξεκινήσει και λειτουργούν καλά, αυτά να μπορέσουν να συνεχιστούν και να πρικοδοτηθούν με τα απαραίτητα κονδύλια. Πολύ καλύτερα λοιπόν να συνεχίσουμε να παραμείνουμε συνεπείς στη γραμμή μας αυτή παρά να καθίσουμε να επινοήσουμε νέα τα οποία σημαίνουν πολλή δουλειά βέβαια, αλλά και κινδυνεύουν μετά να μην μπορέσουν να εφαρμοστούν. Όλες και όλοι οι συνάδελφοι γνωρίζουν ότι για την εφαρμογή των πιλωτικών προγραμμάτων και προπαρασκευαστικών δράσεων, ότι αυτά γίνονται σε πολύ στενή επαφή με τις ε, αρμόδιες υπηρεσίες της Κομισιόν. Δεν χρειάζεται να υπενθυμίσω σε κανέναν ότι το 2014, εάν πρόκειται να ξεκινήσουν νέα προγράμματα, θα εργαστούμε ίσως λίγο μετά το Πάσχα και μετά, για το χρόνο μιλώ και μετά έληξε το κοινοβούλιο όπως έχει σήμερα, μετά, ε, ε, ακολουθεί δηλαδή μετά το Πάσχα του 14 προεκλογική περίοδος, εκλογές και ούτω καθεξής. Άρα, τάσσομαι εδώ υπέρ της ιδέας. Τα χρήματα που διαθέτουμε να τα βάλουμε στα έργα τα οποία ήδη έχουν αρχίσει και όπου ίσως μπορούμε να δώσουμε μια παραπέρα όθηση. Τώρα, οι οργανισμοί μας. Πέντε τον αριθμό, όπως είπε και η Αν Γένσεν. Είναι σημαντικό οι οργανισμοί αυτοί να είναι σε θέση να ολοκληρώσουν την εργασία τους με τους πόρους δηλαδή που θα διαθέτουν, να ολοκληρώσουν τις αποστολές που τους έχουμε αναθέσει. Δεν έχει κανένα νόημα από τις πολλές περικοπές εξοικονομήσεις να περικόψουμε του προϋπολογισμούς των οργανισμών έτσι ώστε στο τέλος να μην μπορούν να αποδώσουν, να μην μπορούν να εκτελέσουν τις αποστολές που του έχουμε αναθέσει. Γνωρίζουμε ότι η Κομισιόν περί τα τέλη του 2011 ανέλαβε την δέσμευση να εξοικονομήσει 5% του συνολικού προσωπικού και αυτό αφορά και τους οργανισμούς. Άρα από το 2012 και για την επόμενη πενταετία κάθε χρόνο να μειώνεται ένα εκατό του προσωπικού. Αυτό ήδη έχει θίξει σοβαρά τους μικρούς οργανισμούς. Και για τους μεγαλύτερους οργανισμούς τίθεται το ερώτημα εφόσον γίνεται αυτό πώς αναθέτουμε και παραπάνω αποστολές. Εγώ είδα πάντως έγγραφο της Κομισιόν όπου λέει ότι πρέπει να γίνουν δραστικές περικοπές και πολύ περισσότερο από μέχρι τώρα. Και όταν γίνονται περικοπές στον ένα, επειδή παίρνουν το συνολικό ποσό όλων των οργανισμών, τότε ίσως μπορούν να δώσουν κάτι παραπάνω σε κάποιον άλλο. Μα δεν είναι πράγματα αυτά. Είναι σαν να πούμε η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος θα λάβει λιγότερα χρήματα και γι' αυτό ίσως δώσουμε ας πούμε περισσότερα στη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης. Αυτά δεν είναι, δεν είναι δυνατόν. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Η Κομισιόν αντέδρασε πάντοτε στο να βάλουμε ξεχωριστή κατηγορία στον προπολογισμό για όλους τους οργανισμούς. Ήθελε πάντα οι οργανισμοί οι οποίοι αποτελούν άλλωστε τμήμα της Ευρωπαϊκής Διοικήσεως πάντα λοιπόν αυτοί να μην μπαίνουν στην κατηγορία 5 αλλά στην εκάστοτε κατηγορία όπου δραστηριοποιούνται. Έφτιαξε λοιπόν γενικές διευθύνσεις εταίρους των οργανισμών αυτών και δεν είναι δυνατόν τώρα να πάρουμε το ψαλιδάκι να κόψουμε λιγάκι από έναν οργανισμό και να το δώσουμε σε άλλον. Κατά τη γνώμη μου πρόκειται για διαδικασία η οποία δεν καλύπτεται. Είναι καθαρά παράνομη. Εφόσον λοιπόν μεμφόμαστε το Συμβούλιο για παράνομες δράσεις, τότε οφείλω να μεμφθώ και την Κομισιόν. Υπάρχει πολλή δουλειά βέβαια και γι' αυτό ο αρμόδιος, οι αρμόδιοι επίτροποι Λεβαντόφσκι και Τσέρτσοβιτ δεν έχουν λάβει καμιά επιστολή ακόμη δική μου. Θα λάβουν όμω και θα έχει το ίδιο αυστηρό ύφο και περιεχόμενο όπω αυτά που σα λέγω τώρα. Να είστε όλοι έτοιμοι για καυγά, διότι δεν μπορούμε να δεχθούμε τέτοια πράγματα που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόεδρο, Γιούτα Χάουκ, ευχαριστώ. Πράγματι βλέπω σε αντιπροσωπείες που μεταβαίνουν στους οργανισμούς αυτούς, του ζητούμε νομοθετικά όλο και περισσότερες αποστολές και δεν μπορούμε τώρα να έρθουμε και να πούμε «Α, σας περικόπτουμε 5%». Υπάρχουν διακυμάνσεις. Εφόσον γίνονται περικοπές, ας κοιτάξει η Κομισιόν τι γίνεται και από τα έσοδα. Δηλαδή, για παράδειγμα, οι κανονισμοί τελών των οργανισμών αν θα πρέπει να τροποποιηθούν. Δηλαδή να μην διοχετεύονται χρήματα στους οργανισμούς, αλλά να φανεί λίγο δημιουργική η Κομισιόν και σε ό,τι αφορά την πλευρά των εσόδων των οργανισμών. Όπως γίνεται και με τους εθνικούς οργανισμούς, ότι δηλαδή αυτοί συγχρηματοδοτούνται από την ίσπραξη εισφορών ή τελών. Αυτή είναι πιστεύω η λύση. Σε ό,τι αφορά τους οργανισμούς, έχω αρκετά εκνευριστεί θα έλεγα σε ό,τι αφορά την απολύτω αδέξια αυτή προσέγγιση τη Κομισιόν. Δεν μπορεί να μεταφερθεί αυτή η περικοπή το 5% έτσι ατόφια στου οργανισμού. Δεν είναι καθόλου τρόπο αυτό. Άλλωστε η κίνηση εκεί δεν είναι κυκλική, είναι όπω είπα ε, περισσότερο μια διακύμανση. Ε, επιθυμούν άλλοι συνάδελφοι να λάβουν το λόγο. Η κυρία Κροστέτ πρώτα. Ε, θα σας ε, θα υποστηρίξω την εισηγητρία μας ε, και συμφωνώ μαζί σας ε, κυρία Ε, Μερικοί από εμά πήγαμε στο Λονδίνο να δουλέψουμε δύο μέρες με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων. Έχουμε την εντύπωση ότι υπάρχει μια αντιπαλότητα μεταξύ των ε, οργανισμών που δημιουργήθηκαν ε, με κατόπιν ετοιμάτων κομισιών, υποστηριζόμενες από το Κοινοβούλιο, ανάμεσα στους οργανισμούς και τις γενικές διευθύνσεις πλέον της Ευρωπαϊκής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και υπάρχει και μια αντιπαλότητα, μια αντισλία ανάμεσα σε νομικούς και επιστήμονες. Και αυτό είναι δυσάρεστο, διότι οι αποφάσεις που οποίες καταλήγουμε τελικά είναι πολύ άσχημες και δεν μπορούμε να τις υποστηρίξουμε. Ας εγγυηθούμε λοιπόν τον προπολογισμό αυτών των υπηρεσιών και των οργανισμών που έχουν πολλή δουλειά να κάνουν. Θα πρέπει να σταθούμε δίπλα τους γιατί αυτό που συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι δυνατόν να γίνει δεκτό. Ευχαριστώ ο κύριος Μπόκρος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. ενδιαφέρουσα η κατάσταση, η εξέλιξη στην Κύπρο, όπου έχει εκπέσει το σχέδιο Α και δεν υπάρχει Β. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και για τον προϋπολογισμό του επομένου έτους, γιατί πρέπει να υπάρχει σχέδιο Β ακόμα και αν δεν έχουμε πολιετές τον ε, Μάιο ή τον Ιούνιο. Θα ήθελα να ρωτήσω την Αν λοιπόν, ποιο είναι το σενάριο το οποίο προβλέπετε τη στιγμή που δεν θα επέλθει συμβιβασμός ε, μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. δεν μπορούμε να, μπορούμε να μιλήσουμε παρά για προέκταση του προϋπολογισμού, παράταση δηλαδή μέσω του πολύετούς. Η χρηματοπιστωτική κρίση έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ποιοτική δουλειά και στην ποιότητα των θεσμικών οργάνων και δεν τους δίνει τη δυνατότητα να βελτιώσουν την εργασία τους. Γιατί σε μια κρίση αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι οι προβλέψεις και ο καλύτερος προγραμματισμός του μέλλοντος. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν την Αν, ποιο είναι το σχέδιο Β. θα είμαστε λειτουργικοί ακόμα και αν δεν εγκριθεί το πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο διότι θα συνεχίσουμε εφαρμόζοντας τον παλαιό προϋπολογισμό. Ίσως πρέπει να γίνει η συζήτηση κάποια στιγμή περιθεσμών και στα Εθνικά Κοινοβούλια. Αλλά να αναλυφθούν χρέη, αυτό είναι αδύνατον. Δεν ξέρω αν στη δική σας χώρα μέλος είναι δυνατόν. Διότι οι απολύπτες όλο και περιμένουν όλο και περισσότερο να λάβουν τα χρήματά τους, διότι έχουμε ένα ολόκληρο κύμα που το σπρώχνουμε μπροστά μας διότι αποφάσισε μεν το Κοινοβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα ότι πρέπει να μπει ένα τέλος σε αυτή την παράνομη κατάσταση. Έρχονται τότε στην εκλογική μας περιφέρεια και μας λένε «Κοιτάξτε, όλο και περισσότερο καθυστερούν τα ευρωπαϊκά χρήματα να μας έρθουν. Έχουμε κάνει για χρηματοδοτήσεις και δεν έρχεται και δεν έρχεται τίποτε». Εγώ βέβαια δεν είμαι εμπειρογνώμων του προπολογισμού. Έτσι λοιπόν θα τηρήσω σιγήν από εδώ και μπρο. αλλά είναι αρκετά, με, αρκετά συναισθηματικά φορτισμένη η ε, υπόθεση αυτή. Η κυρία Γένσεν έχει τώρα πάλι το λόγο ω Γενική Συγκήτρια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας και για την ερώτηση του κυρίου Μπόκρος. Λοιπόν, ε, Σίγουρα, αν δεν καταλήξουμε συμφωνία, δημιουργούνται περιπλοκές. Όμως η συμφωνία αφορά διάφορες, διάφορα επίπεδα. Χρειαζόμαστε συμφωνία για την νομική βάση, χρειαζόμαστε συμφωνία για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αν συμφωνήσουμε την νομική βάση, αλλά όχι το δημοσιονομικό πλαίσιο, έχουμε την οροφή του 2013. Κάτι που δεν είναι πολύ διαφορετικό, αυτή η οροφή, από ε, αυτό που κατέληξαν το αποτέλεσμα των ε, αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων για το 2014. Σημαίνει λιγότερα ποσά για την 1α ε, και για άλλες ε, και για άλλα κονδύλια τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την Επιτροπή σας. Πάντως όλοι θέλουμε να βρούμε λύση και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε επικοδομητικές διαπραγματεύσεις. Αυτή είναι η κατάσταση. Από εδώ ξεκινάμε, αυτό είναι το σημείο εκκίνησης. Τώρα αν χρειαζόμαστε σχέδιο Β. Μερικές φορές ε, δεν πετυχαίνει το σχέδιο Α εκτός και αν γνωρίζει ότι είναι πολύ δύσκολο να καταλήξει σε σχέδιο Β. Τώρα σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς. Ε, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί να εξασφαλίσουμε ότι οι υπηρεσίε οι οποίες έχουν ε, σημαντικό έργο και δουλεύουν καλά θα έχουν επαρκή προπολογισμό. Ε, το, τα προβλήματα προκύπτουν από τους αρχηγούς κρατών κυβερνήσεων οι οποίοι έχουν αποφασίσει συγκεκριμένες ε, ε έδρες για τις υπηρεσίες ε, και αυτό ε, καθιστά δύσκολη τη συγχώνευση υπηρεσιών. Ε, θα μπορούσαν να γίνουν συγχωνεύσεις όχι σε υπηρεσίες της, του δικού σας τομέα υπάρχουν όμως άλλες παλιότερες υπηρεσίες οι οποίες θα μπορούσαν να ε, συγχωνευτούν, αλλά βέβαια αυτό αποφασίζεται από του αρχηγού κρατών κυβερνήσεων. Ε, τώρα, για το τελευταίο από τα σχόλια τη κυρία Γκροστέτ. Ε, τι διαμάχε μεταξύ κομισιών και υπηρεσιών οργανισμών. Νομίζω ότι αυτές θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Γι' αυτό το λόγο το Κοινοβούλιο πρέπει να είναι παρόν να διασφαλίζει ότι ε, οι υπηρεσίες οι οποίες, στις οποίες αναθέτουμε καθήκοντα θα έχουν και τις δυνατότητες να τα εκτελέσουν, να τα φέρουν σε πέρας. Ε, περιμένω όμως με ανυπομονησία να συνεργαστώ με την, Επιτροπή σας όταν μάθουμε περισσότερο, περισσότερο τα δεδομένα στα οποία θα κινηθούν διαπραγματεύσεις. Κύριε Χάουκ, ευχαριστώ. υποστηρίζουμε και νομίζω όλοι την σταθερά βούληση της διαπραγματευτικής μας ομάδας στην οποία νίκη και η Αν Γένσεν όχι υπό την ιδιότητά της ως Γενική Συζήτριας για το 2014 αλλά ως συνεισηγήτριας για τους ιδίους πόρους. Την βούληση λοιπόν όπως είπα να καταλήξουμε σε συμβασμό με το Συμβούλιο για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Από την άλλη πλευρά να μην μας τρομάζει ότι ενδέχεται να μην υπάρξει συμφωνία. Διότι είναι σαφώς ορισμένο το τι θα γίνει σε τέτοιο ενδεχόμενο. Τα είπα, τα έχει πει και η Αν Θα εργαστούμε μετά στη βάση των οροφών που έχουμε ήδη καθορίσει το 2005, με τις οροφές δηλαδή του 2013 όχι με τον πραγματικό προϋπολογισμό του 2013, αλλά με τις οροφές, με τα ανώτατα όρια του 2013, που έχουν γίνει αντικείμενο διαθεσμικής συμφωνίας. Αυτό είναι το πρώτο. Αυτό λοιπόν είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούμε να ε, εγκρίνουμε δαπάνες. Διότι λέει καθαρά στη συνθήκη ότι όλα τα μέχρι τώρα συμφωνηθέντα παραμένουν ως έχουν. Δηλαδή το δημοσιονομικό πλαίσιο, καθώς και η όλη διοργάνωση της συνεργασίας μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Όπως λοιπόν είχαμε αποφασίσει τότε. Σε ό,τι αφορά πολιετή προγράμματα, για παράδειγμα πρόγραμμα δράσεων υγείας και πρόγραμμα LIFE, συμμετέχουμε εμείς με αυτά τα προγράμματα. Εκεί μπορούμε ασφαλώς να συζητήσουμε με τα ειδικά Συμβούλια Υπουργών, ακόμη και αν δεν υπάρχει πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, Εφόσον λοιπόν αυτοί διαθέτουν την πολιτική βούληση, μπορούμε να καθορίσουμε τότε πολιετή προγράμματα. Ασφαλώς, διότι δεν λέει πουθενά η συνθήκη. Το 174 και επόμενα λένε, ναι, λένε κάτι για τα πολιετή προγράμματα, ότι πρέπει να καθορίζει το περιεχόμενο, η διάρκεια τους κλπ. Αλλά δεν λέει τίποτα απολύτως σχετικά με το ότι εξαρτώνται αυτά από πολιτέ σε δημοσιονομικό πλαίσιο. Ε, θα μου πείτε τώρα, μα πώ θα γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Κοιτάξτε, α εξετάσουμε τι κάνουν οι χώρε μέλη. Και εκεί υπάρχουν συνεχιζόμενε πολιτικέ που επαναλαμβάνονται κάθε, χρόνο, κάθε χρόνο και χρηματοδοτήσεις έργων χωρίς σε οποιαδήποτε από τις 27 χώρες μέλη να υπάρχει κάποιο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Υπάρχει απλώς η συνέχιση της πολιτικής. Τα πράγματα δεν είναι διαφορετικά. Εδώ και ο δικός μας προϋπολογισμός βασίζεται στην αρχή της συνέχισης των πολιτικών. Μπορεί λοιπόν, μπορούν να συνεχίζουν τα προγράμματα αυτά και χωρίς πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Άρα δεν δικαιολογείται καμία ανησυχία. το μόνο που θέλω να πω σε όλες και όλους τους συνοδέλφους ότι γίνονται και χωρίς, αλλά βεβαίως είναι πολύ καλύτερα με δημοσιονομικό πλαίσιο. Πρώτα σας ευχαριστώ. Εδώ ολοκληρώνεται η συζήτηση του θέματος και προχωρώ στο επόμενο, τα φθοριούχα αέρια, με εισηγητή τον Μπάς Έικχαουτ, ο οποίος θα κάνει τη σχετική εισαγωγή. Ευχαριστώ και σας ευχαριστώ όλους που παρευρίσκεστε εδώ για αυτό το σημαντικό θέμα. Φαίνεται τεχνική υφής όταν ε, μιλάμε για αυτά τα φθοριούχα αερία, αλλά είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα που αφορά την πράσινη οικονομία. Σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε ε, ότι έχουμε να κάνουμε με φθοριούχα αέρια ε, όπου επιχειρήσεις παραπονούνται ότι θα πτωχεύσουν αν γίνει κάτι. Υπάρχουν όμως και πολλές ε, επιχειρήσεις που ζητούν ενισχυμένη νομοθεσία και εκείνες βεβαίως έχουν επενδύσει σε εναλλακτικές εδώ και δεκαετίες. Και έχει σημασία να δούμε τι θα κάνουμε. Ας αρχίσω με τα φθοριούχα. Πρόκειται για αέρια τα οποία αυξάνουν το δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη μέχρι και 23.000 φορές. Το επίπεδο εκπομπής είναι χαμηλότερο, αλλά η ε, μοριακή τους απόδοση είναι πολύ ψηλότερη. Ε, τα φθοριούχα αέρια επίσης χρησιμοποιούνται στον κλιματισμό, σε εξοπλισμό ψήξης. Μιλάμε για έναν κύκλο ζωής μέχρι 50 χρόνια. Άρα αυτά που θα αποφασίσουμε σήμερα έχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις. Αν δείτε την αύξηση εκπομπών φθορίχων αερίων, βλέπετε ότι είναι ουσιώδης, ιδιαίτερα στα κλιματιστικά. Από το 90 οι εκπομπές αυτές έχουν αυξηθεί κατά 60% και θα αυξηθούν περαιτέρω, γιατί χρησιμοποιούμε όλο ένα και περισσότερο συσκευές κλιματισμού. Άρα θα έχουν ε, ε, δραστικές επιπτώσεις στις κλιματικές αλλαγές, ιδιαίτερα αν δείτε το χάρτη πορείας της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έχουμε λοιπόν μεγάλη αύξηση αν δεν ασχοληθούμε με το θέμα και αυτό μας απασχολεί σήμερα. Θα ήθελα να τονίσω επίσης ότι όταν μιλάμε για φθοριούχα αέρια, μιλάμε για διάφορες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις εντός και εκτός Ευρώπης. Θα ήθελα να τονίσω ότι εάν ρυθμίσουμε καλύτερα, αυτό θα είναι ευεργετικό για την εγχώρια παραγωγή φθοριούχων αερίων και αυτό για την Ευρώπη σημαίνει ε, δράση υπέρ των ΜΜΕ. Όλες οι επιχειρήσεις που παραπονούνται είναι κατά κύριο λόγο αμερικανικές και ιαπωνικές που προβαίνουν σε πολλές εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό θα θέλαμε να υποστηρίξουμε τις ΜΜΕ, τις εγχώριες, τις δικές μας. Ως προς την πρόταση της Επιτροπής, όπως γνωρίζουμε, η Επιτροπή προσπαθεί να βρει μια ισορροπία εντός της Κομισιόν. Υπάρχουν ε, διάφορες δυνάμεις λοιπόν που θέλουν να φτάσουν ε, σε μια πρόταση και ε, διέρευσαν πολλά έγγραφα που ήταν πολύ φιλόδοξα αλλά το τελικό είναι πολύ λιγότερο. Άρα ως εισηγητής στην πρότασή μου προσπαθώ να διορθώσω κατά κάποιο τρόπο αυτή την ε, παλινοδία της Επιτροπής και θέλω να αντιστρέψουμε αυτή την αδύναμη πρόταση. Αν ήμουν ένας πράσινος πολιτικός θα ήμουν ακόμα πιο φιλόδοξος Ξέρω όμως ε, ότι εδώ εκπροσωπώ το Κοινοβούλιο, είμαι εισηγητής του Κοινοβουλίου και θέλω να εξισορροπήσω αυτή την τάση μεταξύ φιλοδοξίας και ευκταίου, ευκταίων στόχων. Άρα θα θέλαμε να δώσουμε μία όθηση στις ΜΜΕ για να δούμε τι εναλλακτικές έχουμε. Μία από αυτές τις ε, εναλλακτικές ε, στα ψυκτικά ε, συστήματα είναι το διοξίδιο του άνθρακα. Αν δείτε, οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα είναι πολύ χαμηλότερες σε σχέση με τα φθοριούχα αέρια. Και υπάρχουν επιχειρήσεις που επενδύουν σε εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Και εξαρτάται από τη ρύθμιση πώς θα εξελιχθεί αυτό το πλαίσιο εκπομπών. Άρα επεκτείναμε τις απαγορεύσεις εκεί όπου υπάρχουν εναλλακτικές. Και στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι να μιλήσουμε για μια φθήνουσα πορεία και απαγόρευση εκεί που χρειάζεται. Δηλαδή, αν συνολικά έχετε το ποσοστό, το ποσό των φθοριούχων αερίων, αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε μία φθήνουσα πορεία στην Ευρώπη, αλλά εάν υπάρχουν εναλλακτικές, θα πρέπει αυτοί οι τομείς να μην φτάσουν σε ενδιάμεσες λύσεις που τρώνε ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της φθήνουσας πορείας. Άρα Όσο περισσότερες απαγορεύσεις υπάρχουν, τόσο μεγαλύτερη ευελιξία θα υπάρχει για προβολή εναλλακτικών λύσεων. Προτείνω λοιπόν απαγορεύσεις σε πολλούς τομείς για να υπάρχει ευελιξία στους τομείς που την χρειάζονται. Προτείνω λοιπόν απαγορεύσεις σε συστήματα ψήξης αλλά και σε μονάδες, σταθερές μονάδες ε, κλιματισμού. Ως προς το, στα συστήματα ψήξης, συναντηθήκαμε τρεις φορές όπου πολλοί εμπειρογνώμονες μας είπαν πως έχει η κατάσταση, οι σκιώδεις παρευρέθηκαν και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για άλλη μια φορά γιατί συμμετείχαν και συνέδραμαν καθώς και φιλοξένησαν αυτές τις ε, συναντήσεις, στα συστήματα ψήξης το θέμα ήταν απόλυτα σαφές. Θα πρέπει η πρόταση να είναι πολύ πιο φιλόδοξη. Ως προς τα ε, μέσα κλιματισμού, εδώ μιλώ για σταθερές μονάδες και κινητές μονάδες κλιματισμού και υπάρχει περιθώριο ευελιξίας γιατί χρησιμοποιήσαμε τις ακροάσεις με τους εμπειρογνώμους για να φτάσουμε σε συμπεράσματα. Ζητώ λοιπόν για, για κλιμακωτή κατάργηση, ιδιαίτερα στον τομέα ψήξης και κλιματισμού. Αυτό μπορεί να γίνει και για έναν άλλο λόγο. Γιατί υπάρχει ένα service ban, δηλαδή σημαίνει ότι η πρόταση της Επιτροπής θεωρεί ότι ως προσορισμένες εφαρμογές θα υπάρξει φθήνουσα χρήση των φθοριούχων αερίων. Σε αυτή τη φάση λοιπόν φθήνουσας πορείας δεν λάβαμε υπόψη το service ban, το οποίο εισήχθη αργότερα, μετά δηλαδή από την φθήνουσα χρήση. Άρα αν χρησιμοποιήσετε το service ban, μπορεί να είστε πιο φιλόδοξοι στην ε, φθήνουσα χρήση αυτών των αερίων. Γι' αυτό θα πρέπει να προλάβουμε τις εξελίξεις και να είμαστε πιο φιλόδοξοι στην ε, φθήνουσα πορεία χρήσης. Επίσης υπάρχει αρχή ορυπαίνων πληρώνει και αυτό σημαίνει ότι αλλάξαμε την πρόταση της Επιτροπής και υπάρχει και ένα εισαγόμενο τέλος, δηλαδή στο τέλος οριπένων πραγματικά ε, καταβάλει αυτό το τέλος για, το για τα φθοριωμένα αέρια θερμοκηπίου και εφαρμόζουμε αυτό το κανονισμό και στις χώρες που πιο δύσκολα μπορεί να εφαρμοστεί διότι υπάρχει διαφορά χρήσης ε, ενδοκινοτικά και υπάρχει ένας διαχωρισμός ε, Νότου και Βορρά. Άρα το σύστημα τελών θα βοηθήσει τις χώρες που έχουν θέματα εφαρμογής πολύ πιο σοβαρά. Άρα δίνουμε μία όθηση στην οικονομία αυτών που επένδυσαν σε ένα φυσικό εναλλακτικό μέσο. Βοηθάμε τις ΜΜΕ μακροχρόνια και προσθέτουμε την αρχή του οριπένων πληρώνει έτσι ώστε να συγκλίνει και το χάσμα μεταξύ Βορρά και Νότου. Αυτά είναι τα θέματα κλειδιά. Θα τα δούμε και με τους σκιώδεις την επόμενη εβδομάδα, να δούμε πώς μπορούμε να φτάσουμε σε τροπολογίες συμβιβασμού. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Μπάς, είναι βέβαια περίπλοκο το θέμα. Έχουμε όμως και άλλη σημαντική έκθεση έτσι λοιπόν προτείνω τρία λεπτά για τους σκιώδεις και δύο λεπτά για τους υπολείπους. Γιατί αλλιώς δεν θα προλάβουμε το άλλο θέμα. Ακολουθεί λοιπόν ο συνάδελφος Μπάνκι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος όπως ζητήσατε. Τρία σχόλια έχω να κάνω. Πρώτον, μικρές κινητές μονάδες κλιματισμού. Από το 2020, σύμφωνα με την πρόταση της Κομισιόν, θα επιβληθεί πλήρης απαγόρευση στην χρήση θρύχων αερίων σε τέτοιου είδους εξοπλισμό. θα χρησιμοποιούνται μόνο φυσικά ψυκτικά. Η προθεσμία 2020 νομίζω ότι είναι πολύ φιλόδοξη. Η, η καινοτομία, μάλλον η, η τεχνολογία, η εναλλακτική τεχνολογία δεν είναι υπό έλεγχο αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή δεν διαφαίνεται η τεχνολογική δυνατότητα να έχουμε αντικαταστήσει τα ε, φθοριούχα αέρια μέχρι το 2020 σε αυτές τις ε, μονάδες. Η Κομισιόν η ίδια δεν ήταν και πολύ σίγουρη αν θα έπρεπε να είναι αυστηρή. Ο εισηγητής από την άλλη μεριά ακολούθησε μια πιο ε, επιθετική πολιτική Ο εισηγητής δηλαδή λέει ότι είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν οι υδροχλωράνθρακες <clears throat> ε, με δυναμικό θέρμανση μεγαλύτερο του 2150. Αλλά είναι προβληματικό για την άποψή μου. Δεύτερον, ε, κινητές μονάδες κλιματισμού στα αυτοκίνητα ε, ε, προθεσμία είναι το 2015 Αν μπορούσατε να μιλάτε λίγο πιο αργά, λέει ο πρόεδρος, διακόπτει τον ομιλητή, ε, για να μεταφράζεστε καλύτερα. Ε, ο κ. Μπάνκη και πάλι, ναι, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, όπως έλεγα, με αυτές τις προθεσμίες. Η έρευνα δεν έχει δώσει επαρκή αποτελέσματα προς το παρόν. Ε, δεν είμαστε σίγουροι ότι τα νέα προϊόντα που έχουν εμφανιστεί με ε, δυναμικό θέρμανση μεταξύ 1 και 20 είναι ασφαλή. Για παράδειγμα σε περίπτωση ατυχήματος όταν διαρρεύσουν από το σύστημα κλιματισμού του αυτοκινήτου. Τέλος, ε, θέλω να μιλήσω για κλιματιστικά σε εμπορικά καταστήματα ε, τι θα γίνει με αυτά, ιδιαίτερα στις χώρες της Μεσογείου. Πρόεδρος, η Γερμανική Ένωση ε, του κλάδου ε, έχει εκδώσει μια ανακοίνωση για το θέμα των κλιματιστικών. Ο κ. Λάινεν. Ε, συγχαρητήρια στον ε, κύριο Άικχαουτ, είναι πολύ προετοιμασμένος ε, και ήταν πολύ χρήσιμες και οι ακροάσεις που έγιναν. Verwendet. Äh, diese Stoffe sind fast überall drin, in allen Kühlgeräten, in allen Klimaanlagen, in äh, Schaltanlagen. Τα φθοριούχα αέρια βρίσκονται σε πάρα πολλές συσκευές κλιματισμού, ψήξης κλπ. κλπ. Οπότε καταλαβαίνετε το ενδιαφέρον του κλάδου. Έχω μιλήσει με πολλούς εκπροσώπους. Τα αέρια αυτά ε, συντείνουν στην αύξηση του φαινομένου θερμοκηπίου. Και θα πρέπει να αποσυρθούν σταδιακά. Υπάρχουν εναλλακτικέ επιλογές, πολύ επαρκείς. Όπως είπα, για τις ψυκτικές εγκαταστάσεις υπάρχουν εναλλακτικέ επιλογές, που κάνουν ένα λόγος να χρησιμοποιούνται αυτοριωμένα αέρια θερμοκηπίου. Πιο δύσκολο είναι για, τις, για τα κλιματιστικά μηχανήματα. Εκεί πρέπει να γίνει κάποια διάκριση μεταξύ τομέων. Εγώ θα προτείνω να εγκύψουμε περισσότερο στην ποικιλία αυτή των μέρων. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατόν να προκύψουν εναλλακτικέ λύσεις, σε άλλες πρέπει να ε, παραταθεί ίσως η περίοδος μετάβασης ή και σε άλλους τομείς δεν υπάρχει και καθόλου εναλλακτική επιλογή. Βέβαια πρέπει να εξεταστούν αυτά, οι εναλλακτικέ επιλογές δηλαδή, και υπό την άποψη της αποδοτικότητας της ενέργειας. Είναι δηλαδή λιγότερη ενέργεια που χρειάζονται αυτές οι εναλλακτικές επιλογές ή είναι περισσότεροι. Χρειάζεται μια συνολική θεώρηση των διαφόρων τομέων. Τώρα, για ψυκτικές εγκαταστάσεις νομίζω μπορεί η ειναι περισσοτερη χρειαζεται μια συνολικη θεωρηση των διαφορων τομεων εκεί να γίνει πολύ γρήγορα. Για τις κλιματιστικές εγκαταστάσεις, όπως είπα, πρέπει να γίνει μια διαφοροποίηση. Νομίζω επίσης πρέπει να υπάρχει και μια απαγόρευση προπλήρωσης των μηχανημάτων. Δηλαδή πρέπει να μπορεί να ελέγχεται στην ίδια την ευρωπαϊκή ζώνη, για εισαγόμενα μηχανήματα δηλαδή, η ε, πλήρωση. Το service ban είναι άλλη υπόθεση τώρα, δεν έχει νόημα μετά από κάποια περίοδο να πληρούνται τα μηχανήματα με ευθοριωμένα αερία Από κάποια στιγμή και μετά πρέπει να πούμε τέλος πρέπει να χρησιμοποιούνται από εδώ και μπρος επιλογές. Κάποιες δυσκολίες αντιμετωπίζω εγώ με τα τέλη που προβλέπει ο Μπάς Eichhout. Για μένα κάτι τέτοιο θα ήταν εφιάλτης να εισπράττονται τέλη οι εισφορές. Ποιος θα τις εισπράττει, ποιος θα τις ανακατανέμει. Αυτό το βρίσκω εξαιρετικά δύσκολο. Εδώ νομίζω ότι υπάρχει αρκετό περιθώριο και ανάγκη συζήτησης. Βέβαια το θέμα είναι σημαντικό και μπορούμε όντω, αν επιτύχουμε κάποια ρύθμιση, να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα στην προστασία του κλίματο. Chris Davis. Δεν είμαι σκιός και προσπαθώ να είμαι και σε δύο επιτροπές ταυτόχρονα. Ε, μιλώ εκ μέρους του κ. Σκυλακάκη. Στην γενική συζήτηση ε, λαμβάνω input και από εταιρείε που λένε ότι είναι πολύ κακή ε, πρόταση και από τον κύριο Έκχαουτ που λέει ότι είναι ακόμα χειρότερη. Ε, όμως ε, άλλες βιομηχανίες του, άλλες εταιρείε του κλάδου ε, είναι πολύ ικανοποιημένες από την πρόταση και λένε ότι θα ε, δημιουργηθούν και καινούργιες ε, ευκαιρίες. με τη μετάβαση σε νέα προϊόντα. Οπότε νομίζω ότι γενικά η Κομισιόν κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ο Μπάς ε, Eckhout ε, έχει υποβάλει προτάσεις που είναι πιο φιλόδοξες από αυτές τις κομισιόν. Μπορούμε να τις δεχτούμε μέσα από αυτές, άλλες είναι πιο προβληματικές. Πάνε πολύ μακριά. Για παράδειγμα, απαγορεύσεις από το 2015 για παράδειγμα μερικών ουσιών. Είναι πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα. Στο μέτρο του δυνατού, θα εξετάσουμε βέβαια τις ε, προτάσεις μία προς μία, δεν έχουμε μία γενική απάντηση. Κάθε πρόταση πρέπει να εξεταστεί διαφορετικά και ξεχωριστά. Η ιδέα σε ό,τι αφορά το service ban ε, είναι καλή για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παρόλο ότι με, με, μερικές μη κυβερνητικέ οργανώσει μιλούν για τη ε, διαφορά μεταξύ βορρά και νότου, θερμοκρασία κλπ. Η αλήθεια είναι ότι θα στοιχήσει περισσότερο στις νότιες χώρες ε, που είναι και πιο φτωχές. Ε, θα είναι πιο δύσκολο να εφαρμοστεί αυτή η νομοθεσία για τα κλιματιστικά από ό,τι στις χώρες του Βορρά. Συνεπώς θα πρέπει να το, να το λάβουμε υπόψη μας. Ε, επίσης το θέμα της προπλήρωσης. Ε, είναι προβληματικό είναι ελκυστικές προτάσει τη Κομισιόν, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την ανάλυση πλήρους κύκλου ζωής. Γεμίζοντας ε, τις συσκευές αυτές ε, από το εργοστάσιο δεν σημαίνει απαραίτητο ότι θα αυξηθεί η εκπομπή ε, ε των σωματιδίων αυτών. Θα είμαστε επικοδομητικοί, θα προσπαθήσουμε να βρούμε καλούς ε, συμβιβασμούς. Ε, χρειαζόμαστε συμβουλές από τους εμπειρογνώμονες, αναθέμα. Δεν ε, θέλουμε να παρασυρθούμε, θέλουμε να λάβουμε, να είμαστε ρεαλιστικοί. Ελπίζουμε ότι θα φτάσουμε πραγματικά σε λογικούς συμβασμούς που θα εξασφαλίσουν την πλειοψηφία και αυτής της Επιτροπής και της Ολομέλειας. Ωραία, λοιπόν, ε, είναι κάτι διαφορετικό αυτό από το να φτιάξουμε ένα ολόκληρο φρούριο από ωραίε πράσινε πέτρε. Η κυρία Γκέρλινγκ. Και εγώ μιλώ εξ ονόματος του Σκιώδους, γι' αυτό θα ήθελα απλώς να μεταφέρω αυτά που έχει να πει ευχαριστή τον Μπάς, τον εισηγητή, Καταρχήν, και τη στιγμή που θα βελτιωθεί η αρχική πρόταση της Κομισιόν υπάρχουν ανησυχίες ως προς την γραμμή μας πλεύσης. Υποστηρίζουμε τις εναλλακτικές ε, υπέρ του περιβάλλοντος και του κλίματος σε σχέση με τα φθοριωμένα αέρια, αλλά δεν θα πρέπει αυτό να σημαίνει φόρτο ως προς τις ΜΜΕ, ως προς την φθήνουσα χρήση, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την χρήση υδροφορανθράκων και δεν θέλουμε να επιταχύνουμε ε, το, την φθήνουσα χρήση πέρα από την πρόταση της Κομισιόν. Γιατί θα πρέπει να δούμε κατά πόσο υπάρχουν τα ποσοτικά δεδομένα για να φτάσουμε τους στόχους ως προς τον έλεγχο της χρήσης άρθρο 1, ως προς την χρήση των φθοριωμένων αερίων, δεν θα θέλαμε να είναι ε, απαρχαιωμένος ο μηχανισμός πριν από το τέλος του κύκλου ζωής του. Και εδώ μιλώ για ε, ψυκτικό εξοπλισμό και κλιματιστικά. Πιστεύουμε ότι χρειάζεται μία εναλλακτική προσέγγιση ως προς την αρχή της απαγόρευσης της, ε, προπλήρωση, της προπλήρωσης θα πρέπει να αυξήσουμε την ενεργειακή απόδοση έτσι ώστε να μην φτάσουμε σε, σε αποτελέσματα τα οποία δεν είναι επιθυμητά. Επίσης δεν θα πρέπει να έχουμε μία γενική προσέγγιση για όλα. Η αρχική απαγόρευση για λόγους ασφαλείας και για λόγους οικονομίας είναι πολύ περιοριστική και αυτό αφορά το παράρτημα. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορούμε να διευρύνουμε το εύρος ε, των απαγορεύσεων. Ως προς τις ε, κατεξιοδότηση πράξης, το θέμα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο. Θα πρέπει να ορίσουμε τις μέγιστες ποσότητες όσον αφορά το παράρτημα 5 και τη χρήση των φθοριωμένων αερίων στην αγορά και θα θέλαμε αυτή η διάταξη να περάσει στο άρθρο 19. Υποστηρίζουμε την πρόταση, θεωρούμε ότι υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης, θα υποβάλουμε τροπολογίες, αλλά θα θέλαμε οι συστάσεις μας να είναι ρεαλιστικές. Äh, ε, κυρία Βίλτς. Εδώ και πολλά χρόνια έχουν αυξηθεί οι εκπομπές των φθοριωμένων αερίων θερμοκηπίου κατά 60% ενώ άλλες έχουν μειωθεί. Άρα εμείς θεωρούμε ότι η πρόταση της Κομισιόν δεν είναι αρκετά, δεν είναι επαρκής. 21% ε, δηλαδή μεταξύ 2008 και 2011 των ε, αερίων που έχουν ε, παραχθεί μπορούν και να απολυθούν. Για να πάρουμε λοιπόν ως βάση για το face down τα έτη 2009 2009-2012, 12. Γινόμαστε γελοί τότε εάν ε, βασιζόμαστε σε απειρχιωμένα νούμερα. Ούτως ή άλλως είναι πολύ υψηλέ οι ποσοστώσεις εάν ακολουθήσουμε την υπόθεση Κομισιόν. Αυτό που χρειάζεται είναι πραγματικές ξεκάθαρες απαγορεύσεις. Για παράδειγμα όπως τα χλώ, στους που επέτρεψε τότε η απαγόρευση εκείνη να προστατευτεί το στρώμα του όζοντος. Η αγορά κυριαρχείται από μια μεγάλη επιχείρηση η οποία θα προσπαθήσει βεβαίως να διατηρήσει την δεσπόζουσα θέση της. Εάν την διατηρήσει όντως, αυτό θα είναι μοιραίο για το περιβάλλον, το οποίο θα συνεχίσει να επιβαρύνεται με αέρια, τα οποία παραμένουν στο περιβάλλον, παραμένουν στην ατμόσφαιρα για δεκαετίες. Υπάρχουν εναλλακτικέ επιλογές που είναι φιλικές στο κλίμα και λιγότερο δαπανηρές. Ορισμένοι θεωρούν ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικέ επιλογές ή ότι είναι πολύ δαπανηρές. Αυτή τη στιγμή όμως η Ένωση επιβάλλει απαγορεύσεις, οι μικρές επιχειρήσεις θα προβούν σε επενδύσεις για να προσαρμόσουν την παραγωγή τους. Οι απαγορεύσεις λοιπόν στην περίπτωση αυτή εξασφαλίζουν και προστασία του περιβάλλοντος αλλά και ασφάλεια σχεδιασμού και είναι επομένω ο μόνο, ο μόνος λογικός δρόμος. Επανέρχομαι στο παράδειγμα των χλωροφθορούχων ε, αερίων που τέλη της δεκαετίας του 80 όλοι είχαν πει τότε οι κατασκευαστές είναι αδύνατο να φτιάξουν ψυγεία χωρίς χλωροφθοράνθρακες γιατί είναι πολύ ακριβά, διότι κτλ. Ωστόσο τα επιχειρήματα αυτά μάλιστα τα ε, επερώνιαν με μελέτες που μετά αποδείχθηκαν εσφαλμένες μετά όμως αναγκάστηκαν να επενδύσουν και όταν οι πρώτοι μικροί κατασκευαστές παρήγαγαν ψυγεία με ε, χρήση εναλλακτικών επιλογών, τότε συνέχισαν και οι άλλοι. Βέβαια, μέχρι να ε, υπάρξουν, να αρχίσουν να χρησιμοποιούνται επιλογές, πρέπει να αποφευθούν ορισμένα πράγματα. Για παράδειγμα, διαρροές διότι οι διαρροές είναι κακές και για το κλίμα και για την, και τσέπη του καταναλωτή. Και επομένως αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Ενάμιση λεπτό δυστυχώ ο καθένα για να μπορέσουμε να συζητήσουμε και την έκθεση τη Λίντα Μακάβαν. Εσείς κύριε Γιούσο. Okay. Θα προσπαθήσω να περιοριστώ στο 1,5 λεπτό. Αυτή η πρόταση κανονισμού είναι καλοδεχούμενη, διότι σε κάθε περίπτωση θα δώσει κίνητρα για επένδυση στην καινοτομία. Καλό και για για τις επιχείρησεις, καλό και για το περιβάλλον. Όμως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τους τομείς και τους κλάδους και που βρίσκονται αυτοί οι κλάδοι. Μιλάμε για πράσινη οικονομία, αλλά ε, μην ξεχνάμε και την πραγματική οικονομία. Η πρόταση λοιπόν είναι καλή, αλλά έχει το άρθρο 11 παράγραφος 3 στο οποίο αναφέρθηκαν και κάποιοι άλλοι που αφορά τον, την απαγόρευση από το 2020 των συσκευών που χρησιμοποιούν αυτά τα αέρια. Να σας μιλήσω για την πραγματική οικονομία. Στη χώρα μου, χώρα του Νότου, ζεστή χώρα, εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν τέτοιου είδου ε, αέρια υπάρχουν πάνω από 4.000. Στην Ολλανδία ούτε καν 150. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. αυτή η απαγόρευση θα σήμαινε αλλαγή της ίδιας εγκατάστασης. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή αέρια εναλλακτικά που να αντικαταστήσουν τα φθοριούχα αέρια. Γι' αυτό μιλώ για την πραγματική οικονομία. Και μην ξεχνάμε και το εξή. Στα ζεστά κλίματα, όπως της χώρας μου, οι, εναλλακτικέ οι εναλλακτικές τεχνολογίες σημαίνουν, συνεπάγονται αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Οπότε, ο τελικός απολογισμός ε, μπορεί να μην είναι και τόσο θετικός που να ε, αξίζει να επιβάλλουμε αυτό το πρόσθετο κόστος επιχειρήσεις. Ας ληφθούν υπόψη οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις λοιπόν. Oui. Πρόεδρε, όπως ξέρετε, η... τα φθορυμένα αέρια ε, μπορούν να βλάψουν 23.000 φορές περισσότερο από το διοξίδιο του άνθρακα από το 90 και μετά, ενώ άλλα τα αέρια θερμοκηπίου έχουν μειωθεί. Ε, μιλάμε για μία ανθυρή αγορά. Το Δεκέμβριο ορίστηκα εισηγητή στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, όπου είμαι αναπληρωματικό, αναπληρωτής. Η έκθεσή μου έχει υποβληθεί για μετάφραση. Θα ήθελα να τονίσω την περιβαλλοντική πτυχή του κειμένου και προτείνω ορισμένες τροπολογίες. Καταρχήν, οι μηχανισμοί πιστοποίησης για το προσωπικό και τις εγκαταστάσεις το 18 και όχι το 15. Επίσης, για την απαγόρευση των φθοριωμένων αερίων θερμοκηπίου τη στιγμή που έχουν, έχουν επίπεδο ε, πάνω από 2.500, δηλαδή μπορούν να βλάψουν και έχουν ισοδύναμο επίπεδο 2.500, να απαγορευτούν επίσης, να απαγορευτούν οι εξοπλισμοί προπλήρωσης ε, πριν από την θέση σε ισχύ του κανονισμού που, προβλέπω το, που εγώ προβλέπω για το 18. Τήρησε το χρόνο μου, δεν μπορείτε να πείτε. Ο κύριος Σπανιό, MEP of the Day. Ζέμπερ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αν θέλουμε να μας πάρουν στα σοβαρά, πρέπει όντως να κάνουμε κάτι στον τομέα των φθοριωμένων αερίων, διότι υπάρχουν μελέτες που δείχνουν τι ζημιά κάνουν. Και νομίζω ότι για την ευρωπαϊκή βιομηχανία ανοίγεται και μια μεγάλη ευκαιρία εδώ να προωθήσει κάποιες εναλλακτικές επιλογές γιατί το θέμα θα γίνεται όλο και πιο σημαντικό. Προβλέψεις της Κομισιόν δείχνουν ότι αν δεν κάνουμε τίποτα το 2050 θα έχουμε τεράστιο ποσοστό εκπομπών αερίων από τα αυτοριωμένα αυτά αέρια. Άρα χρειαζόμαστε κάποιους κάπως πιο φιλόδοξους στόχους. Κατανοώ βέβαια τις ανησυχίες των νότιων χωρών που αντιμετωπίζουν σημαντικότερες προκλήσεις εν προκειμένου. Νομίζω όμως ότι συνήθως υπάρχουν εναλλακτικέ επιλογές και αυτές χρειάζεται να υποστηριχθούν. Και μια φιλόδοξη αντιμετώπιση του θέματος θα εξυπηρετήσει όλους μας και το κλίμα και την βιομηχανία. Και η μακροπρόθεσμη δυνατότητα σχεδιασμού θα πρέπει να είναι στόχος μας. Καινοτομίε και εναλλακτικέ επιλογές. Αυτό που δεν μου φαίνεται σωστό είναι το σύστημα αυτό τελών που προτείνει ο Μπάς Χάουτ. Δεν νομίζω να λειτουργήσει όπως φαντάζεται ο ίδιος. Εγώ θα αποστασιοποιούμουν από εδώ. Προτιμώ να χρησιμοποιήσουμε ρυθμιστικά εργαλεία. Αλλά βέβαια, όπως είπα, με στόχο. Σε Ευχαριστώ. Γκροστέτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα πρέπει να κάνουμε τη διάκριση αφενός του, μεταξύ ψήξης και κλιματισμού. Σε ό,τι αφορά την ψήξη συμφωνώ γενικά. Να σας πω μόνο ότι υπάρχει ένα πρόβλημα της μικρομεσαίας επιχειρήσης γιατί υπάρχει ένα οριακό μέγεθος το οποίο καθορίζει η Κομισιόν. Ίσως θα πρέπει να το ξαναδούμε. Δεν θα πρέπει να πνίξουμε τις μικρομεσίες μας επιχειρήσεις. Μετά, για τον κλιματισμό που είναι κάτι διαφορετικό. Η απαραίτητη τεχνολογία δεν είναι ακόμα διαθέσιμη, δεν έχει αναπτυχθεί. Ε, ίσως δεν θα είναι έτοιμη ούτε πριν από το 2015 ούτε πριν από το 2020. Η Κομισιόν από την άλλη μεριά επιμένει στην προθεσμία του 2020. Μήπως θα έπρεπε, προκειμένου να διαθέτουμε πραγματικά λειτουργικέ αναλυτικέ λύσει, να δώσουμε ε, στου ενδιαφερόμενου άλλα δύο χρόνια, μέχρι το 2022. Σε ό,τι αφορά τι κινητέ μονάδε ε, ψήξη και κλιματισμού, τρένα και αυτοκίνητα, και εκεί δεν έχουμε, μάλλον ούτε εκεί έχουμε ε, την απαραίτητη τεχνολογία. Και στη, τέλος, στην περίπτωση που υπάρχει μια αναλλακτική λύση, σίγουρη, τότε εκεί να είμαστε αυστηροί. Για τις άλλες περιπτώσεις, μήπω θα έπρεπε να δούμε την ημερομηνία, ε, να ξαναδούμε την ημερομηνία 2020 με πολύ κοντά. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, η Κομισιόν, την οποία εκπροσωπεί σήμερα η κυρία Τραμχόρν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Ο στόχος της πρώτης Κομισιόν ήταν να διασφαλίσουμε ότι ο τομέας των φθοριούχων αερίων θα δώσει αυτό που του πρέπει, που του αρμόζει στη μείωση των κομμών δεξιού του ανθρακά. Ε, η έκθεση της 14 Σεπτεμβρίου 2011 του Κοινοβουλίου λέει ακριβώς το ίδιο. Ε, καλεί το Κοινοβούλιο να δράσουμε φιλόδοξα στη μείωση των ε, αερίων του θερμοκηπίου. Αν ε, θέλουμε η πολιτική μας να είναι ευφυή στο μέλλον, δεν θα μειώσουμε απλώς ε, τους, τις εκπομπές, θα αυξήσουμε και την καινοτομία και θα εξασφαλίσουμε πράσινη ανάπτυξη, όπως λέει και ο εισηγητής. Οπότε η Κομισιόν με χαρά βλέπει που η έκθεση, το προσχέδιο έκθεσης του εισηγητή συμφωνεί με τη γενική προσέγγιση που προτείνει η ίδια η Κομισιόν. Σε ό,τι αφορά το επίπεδο της φιλοδοξίας, το βαθμό φιλοδοξίας ε, στην σταδιακή μείωση των εκπομπών, η πρόταση της Κομισιόν βασίστηκε στο πόσο μπορούμε, πόσο μακριά μπορούμε να φτάσουμε με τις υπάρχουσες τεχνολογίες μέχρι το 2000, ε, σήμερα, το 2013. Οπότε, είμαστε σίγουροι ότι τα βήματα τα οποία έχουμε προτείνει είναι εφικτά και έχουμε μάλιστα και περιθώριο ασφάλειας, ιδιαίτερος την πρώτη περίοδο, στην αρχή. Αυτό συνδέεται με το γεγονός ότι στις αρχικές μας ε, προτάσεις, στους αρχικούς μας δεν είχαμε λάβει υπόψη το service ban. Ε, ίσως όμως ένα περιθώριο ασφαλείας είναι χρήσιμο γιατί οι επιχειρήσεις ε, πρέπει να δομήσουν, να διαμορφώσουν τις ε, ε, διαδικασίες παραγωγής τους. Η Κομισιόν θεωρεί ότι η σταδιακή μείωση είναι επαρκής έτσι ώστε να δημιουργήσουν την καινούριες αναλυτικές λύσεις. Πρόσθετες απαγορεύσεις ετέθησαν μόνο εκεί που θέλουμε να αποφύγουμε την παράκαμψη της σταδιακής μείωσης ε, ή εκεί που θέλουμε να καλύψουμε και άλλα αέρια που δεν καλύπτονταν από την σταδιακή μείωση. Οι εμπειρογνώμονες ε, είπαν ότι θα μπορούσαμε να θέσουμε και πρόσθετες απαγορεύσεις σε άλλο τύπου εξοπλισμού, αλλά η Κομισιόν δεν θεώρησε ότι αυτή είναι απαραίτητη για να επιτύχουμε το στόχο μας. Να υπογραμμίσω ότι οι απαγορεύσεις ε, που προτείνει η Κομισιόν είναι εφικτές ε, και σημαντικέ σε ό,τι αφορά το, σχέση κόστος ωφέλους μας. Το ε, επιβεβαιώνουν οι επιρρογνώμονες αυτό. Υπό το φως το ότι επηρεάζονται πολλοί τομείς, πολλοί κλάδοι της οικονομίας, θα ήταν δυνατόν να χορηγήσουμε, μάλλον δεν θα ήταν δυνατόν να χορηγήσουμε ειδικέ παρεκκλήσεις θα πρέπει οι ταυτορούχα αέρια να αντικατασταθούν σχεδόν σε όλες τις εφαρμογές, πρακτικά σε όλες τις εφαρμογές που περιλαμβάνουν τέτοιου αέρια. Ορισμένες από τις προτάσεις του εισηγητή ε, είναι, θα πρέπει να τροποποιηθούν έτσι ώστε να καλύπτουν πραγματικά όλους τους κλάδους. Η Κομισιόν θεωρεί ότι η απαγόρευση προπλήρωση είναι απολύτω απαραίτητη όχι μόνο για να εξασφαλίσουμε τα ωφέλη για το περιβάλλον, αλλά και για να εξασφαλίσουμε θεμητό ανταγωνισμό ανάμεσα στου κατασκευαστέ. Χωρί αυτή την ε, απαγόρευση μπορεί κανείς να εισάγει προϊόντα και εξοπλισμό με φθοριούχα αέρια που δεν θα υπόκεινται στους ίδιους κανόνες που ε, αφορούν ε, την σταδιακή μείωση των εκπομπών και της χρήσης. Ε, μετά έγιναν σχόλια και για το service ban. Το άρθρο δηλαδή 11.3. Καταρχήν να σας πω ότι έχει σχέση μόνο με την ψήξη. Το άρθρο αυτό. Ε, ο... Με τις προτάσεις του εισηγητή δεν μιλούμε για αντικατάσταση εξοπλισμού. Λέμε, όταν γίνεται το πρώτο service θα πρέπει να αντικαθίσταται το αέριο το οποίο περιλαμβάνεται σε αυτή τη συσκευή και έχει GWP 4.000. Ε, Η εναλλακτική λύση έχει ε, δυναμικό θέρμανση περίπου 2.000. Και αυτές οι συσκευές διαραίουν, διαρρέουν τέτοιου είδους αέρια. Ε, σίγουρα λοιπόν καλύτερα να έχουμε ένα αέριο με μικρότερο δυναμικό θέρμανση μέσα. Ε, Επίση, εκφράστηκαν ανησυχίες για το για υπερβολικό άκθος για τις χώρες του Νότου. Αυτό έχει σχέση με την μεγαλύτερη χρήση των κλιματιστικών μηχανημάτων. Γι' αυτό έχω να πω το εξή ότι το συνολικό οικονομικό αντίκτυπος της όλης πρότασης είναι πραγματικά πολύ μικρός. Αν δούμε το έξτρα κόστος του Νότου σε σχέση με το Βορρά εξαιτία της μεγαλύτερης χρήσης συναντιστικών, αυτό φτάνει στο 1 ευρώ κατά κεφαλήν για τις χώρες του Νότου. Αυτό είναι στη χειρότερη περίπτωση, στο χειρότερο σενάριο, διότι οι υπολογισμοί κόστους βασίζονται στις σημερινές τιμές των εναλλακτικών λύσεων. Η... Στην ακρόαση με τους εμπειρογνώμονες ε, που διοργάνωσε ο συγητής μας επιβεβαιώθηκε ότι οι τιμές των εναλλακτικής τεχνολογίας, των εναλλακτικών τεχνολογιών θα πέσουν ε, όταν αρχίσει η ε, παραγωγή τους σε μεγάλη κλίμακα. Αυτή τη στιγμή συγκρίνουμε προϊόντα τα οποία παράγονται σε εκατομμύρια μονάδες με προϊόντα τα οποία παράγονται σε, με, σε εκατοντάδες μονάδες. Συνεπώς, περιμένουμε ότι οι τιμές θα πέσουν και ήδη σε ορισμένα πραγματικά προϊόντα είναι ανταγωνιστικά. Παρακαλώ, ολοκληρώστε, λέει ο Πρόεδρος. Α, είναι δυνατόν, ναι. Ναι, θα ήθελα να πω ότι ε, η, το τέλος είναι κάτι καινούριο. Ε, ε, ας μην αυταπατώμεθα, δεν είναι δυνατόν να ε, αναδιανύμουμε τα τέλη στους τελικούς χρήστες που τα πληρώνουν. Δεν είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Παρακαλώ πάλι σύντομα ο εισηγητής Μπας Έικχαουτ και κυρίως για το σύστημα τελών νομίζω. Α, λοιπόν, μία ώρα μου δίνετε, έτσι δεν είναι πρόεδρε. Όχι, ένα λεπτό μάλλον. Α, δεν άκουσα καλά τότε. Πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, συνεισηγητές μου, Σκιώδης και την Κομισιόν. Και αν μπορώ να συνοψίσω εν συντομία τα όσα άκουσα. Προφανώς υποστηρίζεται την ε, αντικατάσταση στα μηχανήματα ψήξης για τους κλιματισμούς. Ακούω να λέτε ότι πρέπει να διαφοροποιήσουμε αναλόγως με τους διάφορους υποτομείς. Θα είμαι ανοιχτό εκεί σε τροπολογίες, αλλά όσο περισσότερο αρχίζουμε να εγκύπτουμε σε υποτομείς, τόσο πιο πολύ χρειαζόμαστε ορισμούς και ούτω καθεξής. Τέλος πάντων, να ασχοληθούμε με τα θέματα αυτά ε, στον τομέα του κλιματισμού, αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά τους ορισμούς. Για την απαγόρευση προπλήρωσης ακούω πολλούς που υποστηρίζουν ορισμένοι, επικρίνουν, αλλά θέλω να θέσω το θέμα. Δεν έχω ακούσει καμιά πραγματικά ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή για την απαγόρευση προπλήρωσης. Ακούω και, κάποιου και κάποιους που υποστηρίζουν βέβαια. Τώρα, για την απαγόρευση συντήρησης, service ban, άκουσα ορισμένου που αμφιβάλλουν, αλλά νομίζω ότι ο τρόπος που θέτω το θέμα είναι σε μια προσπάθεια να το, κάνω, να το διατυπώσω ακριβέστερα, έτσι ώστε οι απαγορεύσεις συντήρησης να απευθύνονται εκεί όπου πρέπει. Τώρα, για τα τέλη κατανομής, και εδώ είμαι ανοιχτό να συζητήσουμε το θέμα, να συζητήσουμε εναλλακτικέ επιλογές και ούτω καθεξής, αλλά Εν τέλει, και αυτό το έβαλα άλλωστε, υπάρχει ε, μια διαφορά μεταξύ Βορρά και Νότου για το θέμα αυτό. Και το είπαν και ορισμένοι άλλοι συναδελφοί μου. Έτσι λοιπόν ας το δούμε αυτό όταν θα μπούμε στην φάση των ε, τροπολογιών συμβασμού. Ολοκληρώνω εδώ. Δύο λεπτά ίσως είναι κάπως ας πούμε σαν ένα Ολλανδικό λεπτό να το πω έτσι κάπως αυτό που μου ζητήσατε. Ας συνεργαστούμε λοιπόν για να καταλήξουμε σε συμβαστικές τροπολογίες και να μπορέσουμε να προωθήσουμε το θέμα στην τελική έγκριση όσο γίνεται γρηγορότερα. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστώ Προθεσμία καταθέσεως τροπολογιών είναι 28 28η Τρίτου στις 12 το μεσημέρι. Στην Επιτροπή Περιβάλλοντος θα ψηφίσουμε 19 Έκτου και στην Ολομέλεια θα καταλήξει έκθεση, αλλά ακόμα δεν γνωρίζουμε ακριβώς πότε. 28 Τρίτου, 19 ε, Έκτου, όπω είπα, είναι οι δύο ημερομηνίες. Και ακολουθεί το επόμενο θέμα της ημερική διδάξεως, οδηγία για προϊόντα καπνού. Παρακαλώ πρώτα ησυχία και θα δώσω το λόγο πρώτα, κατ' επιθυμία της εισηγητρίας, στην Κομισιόν στον αρμόδιο ε, επικεφαλής μονάδας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ, μην υπερβείτε τα 10 λεπτά. Υπάρχουν πολλοί συναδελφοί μου που επιθυμούν να λάβουν το λόγο, να έχουν λοιπόν την δυνατότητα. Η Κομισιόν. Thank you very much, Mr. President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Εισηγήτρια, αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου, σας ευχαριστώ πολύ που καλέσατε την Επιτροπή σήμερα στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Όπως γνωρίζουμε όλοι, ο καπνός αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκοτώνει 700.000 ανθρώπους ετοσίως, ε, δηλαδή μία πόλη της τάξεως της Φραγκφούρτης ή του Παλέρμο. Μειώνει τη διάρκεια ζωής 50% των χρηστών κατά 14 χρόνια. Αυξάνει τον ε, αριθμό χρόνων ζωής υπό κακές συνθήκες υγείας. Ο έλεγχος λοιπόν χρήσης του ε, καπνού αποτελεί κάτι το ιδιαίτερα επενεταίο αλλά και μια πραγματική οικονομική ανάγκη, αναγκαιότητα. Σας παρακαλώ σταματήστε. Παρακαλώ να πάσουν όλες οι συζητήσεις εντός της αίθουσας και εφόσον επιθυμείτε να συζητήσετε να αποχωρήσετε από την αίθουσα. Όσοι επιθυμούν να ακούσουν τη λέει της Κομισιόν να του επιτρέψουν να μιλήσει μέσα σε ευπρεπές περιβάλλον. Thank uh, Σας ευχαριστώ και πάλι για αυτή την παρένεση. Ε, πιστεύω ότι θα βοηθήσει ιδιαίτερα Άρα πρέπει να αναθεωρηθεί η οδηγία ε, καπνού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οδηγία ήταν του 2001. Θα πρέπει λοιπόν να, και ε, να ενημερωθεί με βάση τις ανάγκες της αγοράς. Θα ήθελα να τονίσω, ιδιαίτερα μιλητής και διακόπτη, Μήπως δεν με ακούσατε και στην τελευταία σειρά, παρακαλώ. Μήπως είναι δυνατόν να σταματήσετε. Θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα την τελευταία πτυχή, την διεθνή πτυχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπογράψει την ε, σύμβαση για τον έλεγχο της χρήσης του καπνού και θα πρέπει νομικά να την εφαρμόσουμε. Επίσης έχουμε δεσμευτεί να ακολουθήσουμε τις κατευθυντήρες γραμμές που ορίζουν τους κανόνες FCT. Βασιζόμαστε στο άρθρο 114 περί ενίας αγοράς και λαμβάνοντας υπόψη ότι ε, λαμβάνουμε υπόψη ότι πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη την αρχή της νομιμότητας καθώς και τις προκλήσεις, θα πρέπει να αρκεστούμε στην εμβέλεια του άρθρου 114. Ήδη μίλησα για τις επιπτώσεις στην υγεία. Με συγχωρείτε, έχασα τις σελίδες μου. Ως προς την ε, ενία αγορά. Μιλάμε για 136 δις ευρώ μετά τέλη. Το 89% αφορά τα τσιγάρα και 7% ε, από τη χρήση καπνού. Στο σχέδιο νέας οδηγίας θα αρκεστούμε σε αυτές τις δύο ομάδες. Μιλάμε για αρχή καπνίσματος, δηλαδή για την αρχή του καπνίσματος που αποτελεί και το μεγάλο όγκο της αγοράς. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις αρχές της αναλογικότητας και να ε, αρκεστούμε στον χαρακτήρα εξισορρόπησης της ε, πρότασης. Μίλησα για τις επιπτώσεις επί της υγείας. Θα ήθελα να τονίσω και ένα άλλο σημαντικό στοιχείο. Το 70% των καπνιστών αρχίζουν πριν από τα 18 τους, 18 τους χρόνια παρά τις προσπάθειες που καταβάλουμε τουλάχιστον να μπορεί κανείς να αγοράσει τσιγάρα μετά από αυτή την ηλικία. Και όταν κανείς φτάσει τα 25, τα 25 του χρόνια, ε, από στατιστικής πλευράς μάλλον δεν θα αρχίσει κανείς να καπνίζει. Γι' αυτό θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στους νέους ανθρώπους. Η πρόταση έχει νόημα και οικονομικά διότι το κόστος ε, υγείας και παραγωγικότητας φτάνει στα έσοδα των ε, βιομηχανιών καπνού, δηλαδή 35 δις. Και είναι συντηρητική η προσέγγιση μας. Γι' αυτό ο πραγματικός έλεγχος ε, χρήσης καπνού είναι κάτι το αυτονόητο. Ας στραφούμε στα βασικά μέτρα. Θα ήθελα να σταθώ σε πέντε τομείς εντάχει. Καταρχήν, συστατικά. Η πρόταση βασίζεται στην χρήση ε, διαφόρων ουσιών flavors, έτσι ώστε να περιοριστούν. Τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να ε, έχουν τη γεύση του καπνού. Θα πρέπει να απαγορευτούν προϊόντα με συγκεκριμένες γεύσεις όπως τεκίλα, σαν αυτό που σας δείχνω. Σήμανση. Δεύτερος μεγάλος τομέας. Προτείνουμε να εισαγάγουμε ε, μια μεγάλη σήμανση προειδοποίησης και στο μπρος μέρος και στο πίσω του πακέτου, δηλαδή το 70% της επιφάνειας να καλύπτεται. Τα κράτη-μέλη μπορούν να ε, καλύψουν και όλη την επιφάνεια δεν θα πρέπει να έχουμε πακέτα σαν αυτά που σας δείχνω, που είναι σαν κραγιόν. Παράνομο εμπόριο, τρίτος τομέας. Θα πρέπει να έχουμε ένα σύστημα ανείχνευσης και χνηλασιμότητας με στοιχεία ασφαλείας για να καταπολεμήσουμε το παράνομο εμπόριο. Τέταρτος τομέας. Ε, σνούς θα πρέπει να απαγορευτεί αυτή η χρήση, δηλαδή προτείνουμε status quo. Πέμπτος τομέας. Ηλεκτρονικά, ηλεκτρικά τσιγάρα που εμπεριέχουν ε, νικοτίνη. Θα πρέπει να αρκεστούμε στην ε, νομοθεσία που ισχύει στον ε, φαρμακευτικό τομέα. Ως προς την εικόνα των νέων πακέτων, έχω ορισμένα πακέτα να σας δείξω. Και πιστεύω ότι στην αποτίμησή μας, στην αξιολόγηση, θα φτάσουμε σε μία μείωση κατανάλωση κατά 2%. Δηλαδή θα σώσουμε τη ζωή 2,5 εκατομμυρίων πολιτών. Αντίθετα, ως προς την καπνοβιομηχανία, τα, οι απώλειες θα είναι, οι ζημίες θα είναι σχετικά χαμηλές και θα πρέπει βεβαίως να λάβουμε υπόψη και την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου. Θα χαθούν 5.000 θέσεις εργασίας, κάτι το οποίο όμως θα αναπληρωθεί με νέες θέσεις εργασίας που θα ανέρχονται στους 8.000. Αυτή ήταν και η παρουσίασή μου, αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο διότι ασχολήθηκε με σπουδή για αυτό το θέμα και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την εισηγήτρια και όλους τους εμπλεκομένους. Σας ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη για τον θόρυβο που με ανάγκασε να σας διακόψω δύο φορές. Ακολουθούμε τώρα, θα ακούσουμε την εισηγήτρια Λίντα Μακάβαν που έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ήθελα να ακούσουμε πρώτα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε να ακούσουν όλοι οι συνάδελφοί μου τι περιέχει η πρόταση και τι δεν περιέχει. Διότι διάφοροι λόμπι, εκπρόσωποι λόμπι θα σας πούνε ότι υπάρχουν πράγματα στην έκθεση τα οποία όμως δεν υπάρχουν. Άκουσα από ορισμένου ότι τα μέτρα α, δεν θα αποδώσουν, δεν θα μειωθεί το κάπνισμα. Από τότε που άρχισαν να λαμβάνονται μέτρα η κυριαρχία του καπνίσματος έχει μειωθεί σε όλες σχεδόν τις χώρες μέλη. Πριν από 50 χρόνια όταν λήφθηκαν στη χώρα μου τα πρώτα μέτρα 70% και 40 ε, των ανδρών και 40 των γυναικών κάπνιζαν. Τώρα έχει μειωθεί ο αριθμός αυτός μετά από μέτρα που έλαβαν οι αρχές. Υπάρχει ωστόσο μια τάση στην Ευρώπη Δηλαδή μειώνεται το κάπνισμα σε όλες τις ομάδες. Σίγουρα ωστόσο ακόμα 29% των νέων καπνίζουν. Δηλαδή μεγαλύτερο ποσοστό κατά μέσον όρο από τις άλλες ηλικιακέ ομάδες. Και από το 2005 και μετά αγόρια από 15 χρόνων ανέρχεται η τάση, δείχνουν τα, τα, τα στοιχεία της ε, Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Αυξάνονται τα ποσοστά αυτά. Δεν θέλουμε να δούμε αντιστροφή τώρα της ε, μειωτικής τάσης. Γι' αυτό συμφωνώ με την Κομισιόν ότι στόχος της νομοθεσίας τους πρέπει να είναι η πρόληψη, η αποτροπή των νέων από το κάπνισμα. Ομάδες λόμπι με τις οποίες έχω συναντηθεί μέχρι τώρα θα σας πούν «Α, ναι, βεβαίως, συμφωνούν με τον στόχο αυτό, δεν θέλουν νεαρούς να βλέπουν να καπνίζουν». Όμως στην αγορά βρίσκουμε προϊόντα σαν αυτό που σας δείχνω, το πακετάκι εδώ, που έχει και η Κομισιόν, κοιτάξτε είναι ροζ, μικρό, χαριτωμένο, έχει ωραία πολύ λεπτά τσιγάρα μέσα, ε, πολύ σικ. Ποιον πάνε να προσελκύσουν με αυτό το design. Στο Στρασβούργο την προηγούμενη εβδομάδα αγόρασα τούτα εδώ. Είναι χαρτιά για να φτιάξετε τσιγάρα με γεύση σοκολάτας. Ποιον πάνε να προσελκύσουν με αυτά. Αυτά πρέπει να ρωτήσουμε μερικού από αυτού του ε, λομπίστε ε, τη ε, βιομηχανία καπνού. Μίλησε η Κομισιόν και για την σύμβαση πλαίσιο που είναι διεθνής και έχει δεσμευτικές διατάξεις και αυτή τη στιγμή εγκρίθηκε και έχει υπογραφεί τώρα από πολλές διαφορετικές χώρες στον κόσμο, οι κυβερνήσεις μας στην Ευρώπη έχουν αρχίσει να την εφαρμόζουν. Έτσι λοιπόν σε διάφορες χώρες της Ένωσης οι κυβερνήσει επιβάλλουν διάφορα μέτρα. Για παράδειγμα, 20 χώρε μέλη έχουν ε, ελάχιστο μέγεθος ε, πακέτων. Έχουμε ε, προειδοποιητικές εικόνες σε ορισμένες χώρες. Άλλες χώρες έχουν λάβει άλλα μέτρα και εθελοντικά μέτρα πέραν της σύμβασης αυτής σε διάφορες χώρες μέλη. Άρα υπάρχουν πολύ διαφορετικά μέτρα. Γι' αυτό κατ' επανάληψη το Κοινοβούλιο στην παρούσα θητεία έχει ζητήσει από την Κομισιόν να υποβάλει πρόταση για τα μέτρα αυτά. Όπως έχουμε ζητήσει και από το Συμβούλιο. Θέλουμε οι κυβερνήσεις να εφαρμόσουν την σύμβαση πλαίσιο όπως την, την έχουν υπογράψει και την έχει υπογράψει και η Ένωση. Βέβαια, η Ένωση πρέπει να πράξει το καθήκον της. Δεν σημαίνει αυτό ότι οι χώρε μέλη δεν πρέπει να κινηθούν προ την διακατεύθυνση. Οι άλλε χώρε. Αυστραλία, το λεγόμενο plain packaging, πακέτα που είναι έτσι. Δεν το βλέπετε ίσως τόσο καλά, αυτό είναι το Αυστραλιανό πακέτο. Και μάλιστα προσέφηγαν στο δικαστήριο κατά της βιομηχανίας και κέρδισαν. Η, το η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου επίσης μιλά για ε, plain packaging και κάτι θα κάνει το Μάη. Άλλες χώρες επίσης προχωρούν σε έλεγχο του καπνού. 63 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο βάζουν προειδοποιητικές εικόνες και 10 χώρες μέλη. Οι Ηνωμένε Πολιτείες έχουν απαγορεύσει τη χρήση ε, διαφόρων γεύσεων εκτός από τη μεντόλη. Το Καναδά το ίδιο. Η Βραζιλία έχει απαγορεύσει οποιαδήποτε χρήση ενισχυτικού γεύσης. Στη Βραζιλία τα ποσοστά των καπνιστών έχουν μειωθεί σημαντικά από 37% σε 15% σε πολλές λατινοαμερικανικές χώρες όπου έχει εφαρμοστεί αυστηρή ε, νομοθεσία καπνού, έχουμε δει να πέφτουν τα ποσοστά των καπνιστών. Σημαντικά. Για τις προτάσεις τώρα. Εγώ θα υποστηρίξω την πρόταση, τις προτάσεις μάλλον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκεί όπου θα προσπαθήσω να τις αλλάξω θα είναι περισσότερο για να τις ενισχύσω. Υποστηρίζω την απαγόρευση των διαφόρων γεύσεων. Γιατί να κάνουμε το κάπνισμα ακόμα πιο ελκυστικό για τους νέους. Το θέλουμε πραγματικά αυτό. Ε, γεύσεις φράουλας, ή Άμα θέλετε πάτε να τα δείτε αυτά τα πράγματα στα καταστήματα στις χώρες σας. Να υποστηρίξουμε λοιπόν την Κομισιόν στην πρότασή της αυτή. Τώρα, συνδυασμός προειδοποιήσεων και εικόνων. Λέει η βιομηχανία ότι αυτά δεν αποδίδουν. Ωστόσο, υπάρχει, υπάρχουν σοβαρέτατες ενδείξεις από τους αρμοδίους. Ρωτήστε και τα Υπουργεία Υγεία σας. Εγώ έλαβα χθε, από ε, Γερμανικό Ινστιτούτο ερευνών ε, καρκίνου που λέει ότι έχουν πραγματικά αποτρεπτική ικανότητα οι ε, εικόνες και οι προειδοποιήσεις για να αποτρέψουν δηλαδή, τους νεαρούς δηλαδή να αρχίσουν το κάψιμα. Η Κομισιόν προτείνει 75% δεν προτείνει το plain packaging, υπάρχει μια διαφορά. Θα βάλουν δηλαδή, θα επιτρέψουν δηλαδή να υπάρχει κάποιο branding, κάποια μάρκα δηλαδή στο τέλος στην Αυστραλία δεν, δεν επιτρέπεται, καν αναφέρεται η μάρκα του, ε, της, ε, του, του τσιγάρου. Για μένα, ωστόσο, αυτό το 75% είναι το απόλυτο μίνιμουμ. Αν θέλουν οι κυβερνήσει να πάνε παραπέρα, να μπορούν να το πράξουν. Εγώ θα ήθελα η Κομισιόν να σχολιάσει, να είναι σαφής δηλαδή ότι αυτή η νομοθεσία, όπως θα είναι, θα επιτρέπει στις χώρες, στις κυβερνήσεις δηλαδή, να πάνε ακόμα περισσότερο, ακόμα μακρύτερα. Θα ακούσετε πολλά από την βιομηχανία που θα λέει ότι τυποποιημένα πακέτα σημαίνουν περισσότερη ε, απάτη, περισσότερες ε, παραποιήσεις. Δεν άκουσα από καμιά δημόσια αρχή όμως να υπάρχουν ενδείξεις για κάτι τέτοιο. Οι δημόσιες αρχές από τις οποίες έχω αντλήσει πληροφορίες, όλες μου λένε ότι δεν είναι δύσκολο να παραποιηθεί ένα από τα τρέχοντα πακέτα τσιγάρων, Πρέπει λοιπόν κάποια ζητήματα να τα πάρετε πολύ σοβαρά υπόψη, γι' αυτό και προτείνουμε ολόκληρη, ολόκληρο τμήμα της προτάσεως σε μια προσπάθεια να ανακοπεί η παραχάραξη, αλλά δεν θα σταματήσει με το να μην βάλουμε πιο μεγάλες προειδοποιήσεις υγείας. Καλύτερα να δούμε τι λένε και οι δημόσιες αρχές για τα πράγματα αυτά. Γιατί άκουσα πολλά τέτοια την προηγούμενη εβδομάδα για το καπνό σνούς. Συμφωνώ με την ε, Κομισιόν. Γνωρίζω ότι ορισμένοι συνάδελφοί μου από την Σουηδία έχουν ανησυχίες. Αν όμως απαγορευτεί στην ευρωπαϊκή αγορά, γιατί να ρυθμίσει ξεχωριστά το σνούς η Κομισιόν. Τώρα, διαμεθοριακές μακρόθεν πωλήσει, δηλαδή μέσω του διαδικτύου. Δεν έχω δει πολλές ενδείξεις νόμιμου εμπορίου διαμεθοριακού. Γιατί να επιτρέπουμε τις ε, αγορές αυτές. Ηλεκτρονικά τσιγάρα τώρα. Αυτά είναι καινούρια προϊόντα στην αγορά μετά από την ισχύ της νέας οδηγίας του 2001. Η Κομισιόν υποβάλλει την πρότασή της που σημαίνει ότι τα περισσότερα ηλεκτρονικά τσιγάρα θα πρέπει να εγκρίνονται ως φάρμακα. Εγώ ζήτησα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναθέσει μελέτη που να συλλέξει όλα τα σχετικά δεδομένα εγώ τίνω να πω μάλλον ότι πρέπει να ρυθμιστούν τα των ηλεκτρονικών σιγάρων. Πολλοί αξιωματούχοι στο τομέα της δημόσιας υγείας θεωρούν ότι ίσως είναι χρήσιμα, βοηθούν ορισμένους να μειώσουν την χρήση των πραγματικών σιγάρων, αλλά πρέπει ωστόσο να έχουν κάποιες, να, να υπακούν σε κάποιες προδιαγραφές. Έχουμε ακούσει κατ' επανάληψη προειδοποιήσει για κινδύνου υγεία από τη χρήση ε, τέτοιων σιγάρων. Ορισμένα περιέχουν περισσότερη νοικοτήνη από ό,τι θα έπρεπε. Οι Ηνωμένε ε, φτιάχνουν δικού τους νόμους τώρα για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, άρα χρειάζεται κάποια ρύθμιση του ηλεκτρονικού τσιγάρου και αναμένω προτάσει για των συναδέλφων. Προβλέπονται πολλέ κατεξουσιοδότηση πράξει μέσα στην πρόταση. Θα τι εξετάσω πολύ προσεκτικά πριν να καταθέσω την δική μου έκθεση για να δω δηλαδή ποιε θα πρέπει να παραμείνουν και ποιε δεν είναι απαραίτητε. Εν τέλει θα σα κάνουν πολύ λόμπι συνάδελφοι, τις επόμενες εβδομάδες για τα πράγματα αυτά. Θα ακούσετε πολλά επιχειρήματα ότι δίθεν οι προειδοποίησει υγείας δεν αποδίδουν, δεν λειτουργούν, ότι οι μεγαλύτερες εικόνες δεν λειτουργούν. Αν όμως όντως δεν αποδίδουν, γιατί έχει λυσάξει το λόμπι απέναντί του. Αν χρειαστεί να πάμε στο δικαστήριο, κοιτάξτε, η καπνοβιομηχανία πάντοτε προσφεύγει στα δικαστήρια. Αν έρθουν να σα πούν κάτι τέτοιο, να είστε βέβαιοι ότι θα προκύψουν δίκες από αυτά τα πράγματα. Η Κομισιόν, ωστόσο, έχει περάσει καιρό πολύ ερευνώντα το θέμα και εμεί πρέπει να τηρήσουμε μια ρωμαλαία στάση. Είναι καθήκον μα να προασπιστούμε του πολίτε, το κοινό. Εγώ δεν θέλω να φύγω από το Κοινοβούλιο του χρόνου τον Απρίλιο όταν θα τελειώσουμε έχοντας το αίσθημα ότι δεν κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να σταματήσουμε αυτή τη νέα γενιά των καπνιστών να, να μην τους αφήσουμε να τους προσελκύσουν οι καπνοβιομηχανίες. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσω με τη συνεργασία σας να καταλήξουμε σε πραγματικά ισχυρά μέτρα ώστε να συνεχιστεί αυτή η τάση μείωση των καπνιστών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Λίντα. Θα διαβάσω τα ονόματα των εγγεγραμμένων. Πρώτα οι Σκιώδη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 Äh, Kabanach, Milan, Pavel Pock, Pilla Ayuso und Sophie Okuni. Habe Μήπως άφησα κάποιο όνομα απ' έξω. Προχωρούμε τώρα στους κύριους ηγητές και δυστυχώς τρίλεπτο. Ή αλλιώς θα αναγκαστώ να μην δώσω το λόγο σε κάποιους που βρίσκονται προς το τέλος του καταλόγου των εγγεγραμμένων. Φλόρεντς, ίσως τα καταφέρω μέσα σε τρία λεπτά, διότι και η Κομισιόνα και η Λίντα είπαν πολλά σημαντικά και δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω. Θα συμφωνήσω σε πολλά με την σοσιαλδημοκράτησα συνάδελφο. Χρειαζόμαστε όντω νέα οδηγία, διότι υπάρχουν πολλά νέα προϊόντα, πολλέ νέε επιστημονικέ ενδείξει και διότι Ε, και διότι έχουμε 300 νεκρούς την ημέρα. Ξέρετε ότι δεν είμαι επιχειρηματίας. Με ενδιαφέρει η διατήρηση της απασχόλησης. Αλλά στη, Γερμανία, στη γερμανική καπνοβιομηχανία έχουμε 6.000 εργαζόμενους. Αλλά για διαιρέστε το με τους 300 νεκρούς, σε 20 μέρες έχουμε καθαρίσει. Ε, είναι σαν να πέσουν αντίστοιχα αεροπλάνα με 300 επιβάτες, κάθε μέρα ένα. Ε, θα διακόψουμε αμέσως τις αεροπορικές συγκοινωνίες. Έχουμε ξεχάσει τι καημό, τι πόνο, τι δάκρυα προκαλούν αυτά τα πράγματα όταν πεθαίνουν οι άνθρωποι από το κάπνισμα νομίζω ότι οφείλουμε να κινηθούμε. Γι' αυτό λοιπόν τα οικονομικά κριτήρια για μένα δεν είναι τόσο πολύ στο προσκήνιο όσο λένε ορισμένοι. Είναι κάπως μακάβριο το επιχείρημα. Ε, πεθαίνουν 7.000 άνθρωποι το χρόνο. Α, ε, να, γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται διαφήμιση, γιατί πρέπει τα χιλιάδες καινούριου πελάτες. Όποιος εξετάσει ρεαλιστικά τις ενδείξεις ωστόσο θα δει ότι με αυτά τα νέα τσιγάρα, κυρίως αυτά τα λεπτά, υπάρχει ανωδική τάση. Μιλώ διότι γνωρίζω για τους νέους και τα δικά μου τα παιδιά δυστυχώς δεν είναι τόσο τέλεια όσο θα ήθελα. Έχουν δίκιο λοιπόν και η Λίντα και η Κομισιόν. Μπορεί κανείς να διαφωνήσει για το εάν οι εικόνες πάνω στα πακέτα θα πρέπει να καλύπτουν το 70% ή το 75%. Αλλά και οι γιατροί ακόμη λένε ότι χρειάζεται να υπάρξει προειδοποίηση, κυρίως για τους νέους, το πόσο επικίνδυνα είναι τα τσιγάρα. Για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα δεν θα τοποθετηθώ σήμερα. Υπάρχουν επιχειρήματα ενδιαφέροντα και από τις δύο πλευρές. Χρειάζομαι κάποιο χρόνο για να μπορώ να πω κάτι με κάποια βάση, ας το πω έτσι. Ακούω επίσης, πού βρίσκομαι τώρα, α, ακούω περί πειρατείας. Αγαπητή καπνοβιομηχανία, τα έχουμε εξετάσει τα πράγματα αυτά. Τα μισά από τα παράνομα τσιγάρα προέρχονται από δική σας παραγωγή. Μέγα μέρος της παραγωγής σας φεύγει από τα εργοστάσια σας και πηγαίνει και λαμβάνει παράνομες οδούς και άτραπους. Φρέντερικ. Φρέντερικ μάλλον. Θα μιλήσω εν συντομία, τα βασικά σημεία, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Καταρχήν συμφωνώ με τον ε, εισηγητή και τον σκιώδη εισηγητή του ΕΛΚ. Είναι τα γνωστά επιχειρήματα τα οποία μας αντιπαραθέτουν, ε, για παράδειγμα, της θέσης ρασίας που κινδυνεύουν, ε, οι, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλπ. Ε, τα στατιστικά όμως που υπάρχουν για τους θανάτους στην Ευρώπη είναι πολύ πιο ισχυρά. Ε, μετά να κάνουμε λιγότερο ελκυστικό τον καπνό για τους νέους, συμφωνώ. Δεύτε, μετά, για, τις, για τη συσκευασία υπάρχουν διαφορετικές ε, θέσεις, σκέψεις και θέσεις, αλλά συμφωνώ με την Κομισιόν. Ε, συνδυασμό εικόνας με κείμενο στο 75% της επιφάνειας του πακέτου. Τώρα βέβαια σε τι αναφέρεται και στις δύο πλευρές ή μόνο στη μία. Ε, ε, γίνεται πρόοδο σε σχέση με το σημερινό καθεστώς. Ε, ζητώ συγγνώμη που μιλάω γρήγορα, λέει η κυρία Σε ό,τι αφορά τα χρώματα και τα πρόσθετα τα, και επίσης τα, τα αρώματα, νομίζω ότι είναι μια πρόταση απολύτως απαραίτητη, κλειδί, πολύ σημαντική γιατί γνωρίζουμε στατιστικά ότι ένας από τους παράγοντες που καθιστά ελκυστικό το κάπνισμα ε, είναι αυτός, αυτές οι ουσίες. Ε, χρησιμοποιούν αυτή τη φλέβα χρυσού, αν θέλετε να το πω έτσι, οι καπνοβιομηχανίες για να προωθήσουν τα τσιγάρα τους, ε, τα προϊόντα τους. Μετά θα πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί με τα προϊόντα καπνού τα οποία πιο πολύ πολλούνται, το καπνό για στρεφτά τσιγάρα, τα τσιγάρα βέβαια. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με την εξαίρεση για τα ε, προϊόντα τύπου για καπνό, για πίπα, πουρα κλπ. Ε, για τα σιγαρίλο ε, θα είχα να πω κάτι. Υπάρχουν στατιστικές από τον Καναδά που λένε ότι αυτά τα αρωματικά τσιγάρα είναι πολύ ελκυστικά για τους νέους. Αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία όλο και περισσότεροι, πολύ μικροί νέοι, μεταξύ 6 και 12 ετών, τα καταναλώνουν. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τα συγκαρίου, λοιπόν, τα αρωματικά τσιγάρα. Τώρα, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, πολύ σημαντικά, δεν μιλούσαμε για αυτά πριν από 10 χρόνια, δεν υπήρχαν τότε. Όμως η εκρονοβιομηχανία καινοτομή. Ε, πιστεύω ότι η Κομισιόν είναι λίγο υπερβολικά αυστηρή με το άρθρο 18 είναι σημαντικό ασφαλώς να εξασφαλίσουμε ότι είναι ασφαλή οι δόσει κλπ. Ε, αλλά ας είμαστε και πιο ρεαλιστές, ας εξετάσουμε τα όρια. Ε, τελειώνω πρόεδρε. Θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστικοί ε, και κυρίως ε, να έχουμε επιχειρήματα εναντίον το αντιεπιχειρημάτων εναντίον των επιχειρημάτων της ε, καπνοβιομηχανίας υπέρ των ηλεκτρονικών τσιγάρων. Ευχαριστώ. Good. Χάση. Ευχαριστώ πολύ. Η εισηγήτρια, η κυρία Μακάβεν, μου καθιστά το έργο ευκολότερο γιατί υποστήριζω επί της ουσίας όλα τα θέματα που Έφυξε η πρόταση της Επιτροπής είναι ευπρόσδεκτη, είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και θεωρούμε εδώ στο Κοινοβούλιο ότι πρέπει μόνο να βάλουμε κάποια τάξη στην αρχική αυτή πρόταση της Κομισιόν. Από την πλευρά των πρασίνων θα θέλαμε στην οδηγία να εισαχθεί ε, αυτό ακριβώς που υπάρχει στην Αυστραλία, δηλαδή ένα απλό πακέτο, plain packaging, όπου δεν φαίνεται η μάρκα. Στην Αυστραλία αυτό ήδη ισχύει. Πολλοί συνάδελφοι τόνισαν ότι θα πρέπει να ασκήσουμε πρόληψη περισσότερο, δηλαδή να προλάβουμε τους νέους από το να αρχίσουν το κάπνισμα. Αν ένα 94% των καπνιστών αρχίζουν πριν από τα 25 και 70% κάτω από τα 18, τότε θα πρέπει να προβούμε σε μία άλλη στοχοθέτηση της αγοράς δηλαδή να προλάβουμε τους νέους ως προς την απαγόρευση των ε, ενισχυτικών ουσιών γεύσεων, θα θέλαμε να επεκταθεί αυτή η απαγόρευση, όχι δηλαδή μόνο αυτό που προανέφερε η Επιτροπή, ε, όχι μόνο να μιλάμε για χαρακτηριστικά αρώματα, αλλά να απαγορεύσουμε όλες τις ε, γεύσεις και τα αρώματα. Αυτό αφορά και τις διαφημίσεις στα σημεία αγοράς. Θεωρούμε ότι τα προϊόντα καπνού δεν θα πρέπει να είναι τόσο ορατά εκεί όπου πολλούνται και ίσως αυτό να οθούσε σε μία μείωση των πωλήσεων. Και έχουμε παραδείγματα προς ε, κάτι τέτοιο, προς αυτή την κατεύθυνση. Όταν οι άνθρωποι δεν βλέπουν κάτι, δεν έχουν και το κίνητρο πάντα ε, αυτή την πρωταρχική όθηση να αγοράσουν κάτι. Έχω λάβει πολλά ε, mail από τα lobby για τα ε, e-cigarettes και αυτό που έχει σημασία είναι να φτάσουμε σε μία εξισορρόπηση τα ηλεκτρονικά τσιγάρα θα πρέπει να αποτελούν μέσο στήριξης για να σταματήσει κανείς το κάπνισμα, αλλά δεν θα πρέπει να αποτελέσουν ένα νέο ε, ε, διάβλο χρήσης και έθισης, εθισμού στην νοικοτήνη. Θα πρέπει να υπάρχει ένα όριο ως προς την ε, χρήση νοικοτήνης στα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Ευχαριστώ πολύ, λέει ε, η κυρία Ρόσμπαχ. Θεωρώ, όπως είπε και η Κομισιόν, ότι καταρχήν θα πρέπει να αναχαιτήσουμε τους νέους έτσι ώστε να μην καπνίζουν. Θα πρέπει να εκπονήσουμε ε, μία μεθοδολογία που να δείξει τους νέους ότι δεν είναι και τόσο ωραίο, δεν είναι και τόσο cool να καπνίζουν. Η Λίντα έχει απόλυτο δίκιο. Γιατί μας λένε ε, δύο διαφορετικά πράγματα από την βιομηχανία. Εδώ δεν μιλάμε για στοχοθέτηση ενός κοινού ενηλίκων όταν έχουμε αρώματα σοκολάτας, γεύση σοκολάτας για να στρίβει κανείς τσιγάρα και ούτω καθεξής. Η στοχοθέτηση είναι συγκεκριμένη. Ξέρουμε ότι ο καπνός βλάπτει την υγεία, αυτό το ξέρουμε όλοι. Αλλά θέλει η βιομηχανία να το ε, προωθήσει σαν χόμπι, σαν πηγή χαράς, όπως όταν πίνει κανείς ένα ποτήρι ουίσκι. Γι' αυτό θα πρέπει να αποτρέψουμε τους νέους. Εάν απαγορευτούν οι διαφημίσεις, πρωτίστως, και αν ε, μία καπνοβιομηχανία δεν μπορεί να δείξει τα προϊόντα της, μας προβάλλουν ότι πρόκειται για στρέβλωση ανταγωνισμού. Εμείς επιδοτούμε τα καπνά και την καπνοκαλλιέργεια στην Ευρώπη. Η καλλιέργεια καπνού επιδοτείται στην Ευρώπη και θα πρέπει να σταματήσει. Γιατί το σναφ τα τσιγάρα και τα συγκαρίγιος ε, την χάνουν της ίδιας αντιμετώπισης. Τα πουράκια. Γιατί υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση. Γιατί αν μιλάμε μόνο για τα πουρα και τα πουράκια, τα οποία ε, παρασκευάζονται με καπνά, κανένας δεν μπορεί να καπνίσει 20 ή 40 την ημέρα. Τουλάχιστον τα 12 χρόνια δεν μπορούν. Άρα η Λίντα έχει απόλυτο δίκιο η βιομηχανία μας λέει δύο διαφορετικά πράγματα. Μιλάει με ε, αυτή τη διπλή γλώσσα και θα πρέπει να σταματήσουμε με τα επωνομαζόμενα candy cigarettes. Δηλαδή να απαγορεύσουμε αυτές τις προσθετικές ουσίες που καθιστούν τα τσιγάρα πολύ πιο ελκυστικά. Γιατί δεν έχουν και την ίδια κατανάλωση όπως έχουν τα πουρα και τα ποράκια. Ευχαριστώ κυρία Ρόσπαχ, η κυρία Άντερσον. Η αρχική μου αντίδραση είναι ότι είναι η... Είναι στη σωστή, ότι η προτάσει είναι σωστή κατεύθυνση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ευθύνη να κάνει τα βήματα που χρειάζονται για να εδραιώσει τα θετικά αποτελέσματα που έχει δώσει οδηγία προεδρών καπνού, ιδιαίτερα για το ακροτήριο των νέων ανθρώπων. Θα πηγαίνουμε ε, ακόμα πιο μακριά μάλιστα. Οι προτάσει Κομισιόν για υποχρεωτική αφαίρεση του 75% της επιφάνειας των πακέτων να καλύπτονται με εικόνες και κείμενα προειδοποιητικά είναι σωστή, αλλά λυπάμαι που δεν πάει ακόμα πιο μακριά να δεν ακολουθεί το Αυστραλιανό παράδειγμα. Θα πιέσω για πιο φιλόδοξη λύση, όχι στο 100% βέβαια που δεν είναι εφικτό, αλλά πιο φιλόδοξο, κάτι πιο φιλόδοξο. Σε ό,τι αφορά τα αρώματα και τα πρόσθετα, ε, η πρόταση της ε, Κομισιόν για το κατά πόσον ε, για τη δημιουργία πάνελς είναι ανέφικτη, είναι γραφειοκρατική πιστεύω θα πρέπει να πάμε πιο μακριά. Να απαγορεύσουμε όλα τα πρόσθετα και αρωματικά και τις αρωματικές ύλες. Οποιοδήποτε οτιδήποτε υλικό δεν χρειάζεται απαραίτητο για την κατασκευή του τσιγάρου, αλλά ελκύει περισσότερο τους καπνιστές, ε, πιστεύω θα πρέπει να απαγορευτεί, ε, γιατί με αυτόν τον τρόπο ε, αυξάνει τον αριθμό των καπνιστών ή διατηρεί, ε, προσελκύει τους ε, περισσότερους καπνιστές. Σε ό,τι αφορά τις διασυνορικές ε, πωλήσει εξ αποστάσεως, θα πρέπει να απαγορευτούν. Θα ήταν κάτι πιο απλό από το σημερινό κείμενο. Γιατί αυτή τη στιγμή θα πρέπει να εφαρμοστούν συστήματα προσαρμοσμένα σε Δεν το κατάλαβα πώ θα λειτουργούσαν κάτι τέτοιο. Το καπνό είναι ένα νέο προϊόν και έτσι θα πρέπει να του συμπεριφερθούμε. Σε ό,τι αφορά το θέμα των ηλεκτρονικών τσιγάρων που άρχισε να καπαρώνει συζήτηση. Δεν πιστεύω ότι ο κανονισμός, ο γενικός κανονισμός προϊόντων δηλαδή είναι επαρκής. Ε, έχουμε ε, δει παραπλανητική σήμανση ηλεκτρονικών τσιγάρων. Ο κανονισμός περί φαρμάκων θα εξασφάλιζε ότι αυτά τα προϊόντα θα έχουν επαρκή ποιότητα, θα είναι ασφαλή και θα αποφύγουμε να απολούνται ή να προωθούνται σε νέους και παιδιά. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι ό,τι κυκλοφορεί στην αγορά θα είναι ασφαλές αν χρησιμοποιείται με το σωστό τρόπο. Και οι χρήστες θα πρέπει να γνωρίζουν τους κινδύνους, ε, ιδιαίτερα αν τα ηλεκτρονικά τσιγάρα αφαιθούν ελεύθερα στα χέρια των παιδιών. Εκεί μπορεί να ε, είναι θανατηφόρα μάλιστα. Λυπάμαι επίσης που δεν αναφέρονται ε, περιορισμοί για τις διαφημίσεις στα σημεία πώλησης. Ε, αναφέρθηκε αυτό από έναν από τους ευρωβουλευτές. Ο πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια δύο, δύο δευτερόλεπτα πρόεδρε στην Ιρλανδία. Ε, όταν κρύψαμε τα προϊόντα καπνού στα σημεία πώλησης ε, είδαμε σημαντική μείωση της κατανάλωση. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ε, παρακαλώ πολύ σεβαστείτε το χρόνο σας ο καθένας, αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να τελειώσουμε. Κλαίνεις. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να έχουμε plain packaging, να μην αναφέρονται οι μάρκες και να απομακρύνουμε τις αρωματικές ουσίες και τις γεύσεις. Θεωρείται ένα προϊόν υπέρ του καταναλωτή και τη στιγμή που υπάρχει υψηλό ποσοστό εθισμού δεν καταλαβαίνω γιατί δεν υπάρχει ρύθμιση ε, πολύ περισσότερα από άλλα απλά είδη όπως το στυλό που κρατώ οι Ευρωπαίοι καταναλωτές θέλουν να δοκιμάζονται τα προϊόντα, τους, τα προϊόντα πριν μπουν στην αγορά. Γι' αυτό θα πρέπει να ρυθμίσουμε και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα θα πρέπει να θεωρηθούν φαρμακευτικό σκεύασμα έτσι ώστε να βοηθούν τον καπνιστή να σταματήσει το κάπνισμα. Είναι πολύ ανησυχητικό το πώς τίθενται σε εμπορία και πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να τα τυποποιήσουμε. Εάν τα τσιγάρα αυτά βοηθούν για, το, για να σταματήσει κανείς να καπνίζει, ε, θαυμάσια. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε κατά πόσο λειτουργούν όπως τα έμπλαστρα, όπως οι τσίχλες και ούτω καθεξής. Δεν πρέπει να αφήνουμε παραθυράκια. Ρεμπέκα Τέιλερ. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με την εισηγήτρια και άλλους συναδέλφους που μίλησαν σχετικά με τις αλλαγές στα πακέτα και στις ετικέτες. Διερωτώ όμως ωστόσο γιατί υπάρχει στην πρόταση και κάτι το οποίο απαγορεύει τα composite cans, δυστυχώς η δεν ξέρει τι είναι αυτό, και ίσως θα έπρεπε κάποια από αυτά να επιτρέπονται. Τώρα, για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα που περιέχουν δηλαδή νικοτίνη, Υπάρχουν ενδείξεις από το ε, Εθνικό Ινστιτούτο Καπνού στην, ε, στην, στο ε, Ηνωμένο Βασίλειο και από άλλους οργανισμούς ότι μπορούν όντως να συμβάλλουν στην μείωση του αριθμού των καπνιστών. Πρέπει να διασφαλίσουμε βέβαια ότι τα προϊόντα αυτά δεν θα είναι ελκυστικά σε μη καπνιστές, να μην ομαλοποιήσουμε το κάπνισμα, να δούμε τις διαφημίσεις και ίσως οι ε, κυβερνήσεις θέλουν και να απαγορεύσουν και τις σχετικές διαφημίσεις. Και βέβαια και επιβολή ορίου ηλικίας για την προμήθεια αυτών των ηλεκτρονικών σιγαρέτων. Επίσης να μπουν πάνω και προειδοποιήσεις που να λένε προσοχή βλάπτουν την υγεία. Αλλά βέβαια δεν είμαστε ακόμα σίγουροι γι' αυτό. Σόνικ, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι το οποίο δεν έχουμε σχολιάσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα όριο σε ό,τι αφορά το πάχος τη διάμετρο δηλαδή του τσιγάρου. Γιατί μόνο στη διάμετρο και όχι στο μήκος, ρωτά κάποιος, κανείς. Ε, τέτοιου είδους ε, προτάσεις είναι τροφή σε αυτούς που προσπαθούν να γελιοποιήσουν ε, την, ε, τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα λένε ότι προσπαθούσαμε να επιβάλλουμε μέτρα για την καμπύλη μιας μπανάνας. Κάτι παρόμοιο, κάπως έτσι ακούγεται και αυτό. Τώρα, έχω τις εξής προς την Κομισιόν. Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν να διατηρήσουν τα τσιγάρα μεντόλ ε, χωρίς ε, τους περισμούς που έχουν υποβληθεί στα, στα άλλα τύπου, στους άλλους τύπους τσιγάρων. Μήπως πρέπει να το δούμε κι εμείς αυτό. Τρίτον, η Κομισιόν είπε πως θα προτείνει νέες μεθόδους για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου, του λαθρεμπορίου τσιγάρων. Μπορεί να μας εξηγήσει. Πέτερ Λίζε, ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ Και Πρόεδρε, ευχαριστώ την Λίντα Μακάβαν και τον Καλάιτ Φλόρεντς του Λαϊκού Κόμματος. Εγώ υποστηρίζω κατά βάση την πρόταση της Κομισιόν Νομίζω βέβαια ότι χρειάζεται να ρυθμιστούν ακόμη και κάποια λεπτομέρειε, δηλαδή στάνταρτ μέγεθος πακέτου, δεν ξέρω αν είναι αυτό απαραίτητο, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται έτσι, πάρα πολύ έντονες ε, ε απαγορεύσεις. Δεν νομίζω θα μπορέσουμε τελικά να απαγορεύσουμε το κάπνισμα ούτε και από την πίσω πόρτα. Χρειάζεται οι καπνιστές βοήθεια για να ξεφύγουν από το κάπνισμα. Χρειάζεται κάποια ρύθμιση και πρέπει να βρεθεί η σωστή λύση για τις επιδοτήσεις, συμφωνώ με την Άννα Ρόσπαχ. Δεν το έχουν προσέξει όλοι. Το Κοινοβούλιο αποφάσισε, διακόπτει ο Πρόεδρος. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την Ιταλική διερμηνία. Βέβαια δεν βλέπω να υπάρχουν Ιταλοί συνάδελφοι, αλλά δεν, υπάρχουν, δεν υπάρχει Ιταλική μετάφραση. Είναι αλήθεια αυτό που λέω. Καλά δεν υπάρχουν Ιταλοί εδώ. Ωραία, συνεχίζουμε χωρίς τα Ιταλικά, τι να πω. Ε, οι Ιταλοί λομπίστες καταλαβαίνουν αγγλικά, συνεχίζω. Όμως να, να μου δώσετε τα έξτρα δευτερόλεπτα που μου πήρατε. Ξανάρχομαι λοιπόν στις επιδοτήσεις καπνού. Ίσως να μην το παρακολουθήσατε όλοι. Δυστυχώς την προηγούμενη εβδομάδα το Κοινοβούλιο αποφάσισε να επαναφέρει τις επιδοτήσεις προϊόντων καπνού. Ελπίζω το Συμβούλιο να μην το επιτρέψει. Το πιο σημαντικό που θέλω να πω είναι η προστασία απέναντι στο παθητικό κάπνισμα. Εδώ μπορεί να βελτιωθεί η πρόταση της Κομισιόν, διότι οι διάφορες προειδοποιήσεις που μελετούμε και θα μπουν και στην επιτροπολογία κτλ. απευθύνονται κυρίως στους ίδιους τους καπνιστές και στον κίνδυνο που αποτελεί το κάπνισμα για τη δική τους υγεία. Αυτό είναι σημαντικό, βέβαια, ιδίω για τους νέους. Αλλά ακόμα πιο σημαντικός είναι ο κίνδυνος για τους τρίτους και ιδίω για τα παιδιά. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα από διάφορες χώρες. Α, όχι κύριε Πρόεδρε, με επιτρέψετε να ολοκληρώσω γιατί με διακόψατε προηγουμένως. Υπάρχει λοιπόν, ε, υπάρχουν λοιπόν πρόοροι τοκετοί, υπάρχουν επίσης πρόοροι θάνατοι, ευνίδιοι θάνατοι βρεφών που οφείλονται στο κάπνισμα τρίτων προσώπων. Τώρα, Παρβάνοβα. 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα πρέπει να σας πω ότι εδώ πρόκειται για σύγκρουση συμφερόντων. Εγώ είμαι γιατρός και θα ήθελα να πω ότι αντιτάσσουμε στη χρήση καπνού, δημιουργεί προβλήματα υγείας, πρόορους θανάτους και ούτω καθεξής. Και νομίζω ότι αν ε, υπάρχουν συνάδελφοι που θέλουν ότι προστατεύουν τους ε, καπνοκαλλιεργητές, τους εργαζόμενους και ούτω καθεξής, θα ήθελα να μιλήσουμε για περίπτωση σύγκρουση συμφερόντων. Υποστηρίζω τη Λίντα Μακέιβον και την Κομισιόν γιατί θέλουμε να μειώσουμε τους καπνιστές κατά 2% και να ε, περισσώσουμε 2,5 ε, εκατομμύρια ζωές τα επόμενα χρόνια. Δεν ξέρω ε, αν κάτι αξίζει περισσότερο από αυτό. Η Λίντα μας έδειξε στοιχεία που δείχνουν ότι η καπνοβιομηχανία δεν θέλει να συνεργαστεί. Θέλει να δελεάσει τους νέους και δημιουργεί κέρδη για τους μετόχους και για τη βιομηχανία. Αυτό θέλουμε να καταπολεμήσουμε και τα λόμπι που περιστρέφονται εδώ γύρω-γύρω και προσπαθούν να μας προσελκύσουν. Εάν θεωρήσουν ότι τα μέτρα αυτά δεν είναι αποδοτικά, θα πρέπει να ζητήσουν ακόμα πιο περισταλτικά ε, νέα ε, μέτρα, έτσι ώστε να μειώσουμε το κάπνισμα κατά 2% και να περισσώσουμε 2,5 εκατομμύρια ζωές. Ευχαριστώ. Να υποφεληθώ της ευκαιρίας για να στηρίξω τις ε, προτάσεις ε, της Κομισιόν και της Ισχύτριας Είναι ένα θέμα δημόσιας υγείας. Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες μας είναι στο επίκεντρο. Είναι μια πρόταση που περιμέναμε εδώ και πολύ καιρό. Συμφωνώ ότι το, ο καπνός θα πρέπει να φαίνεται σαν καπνός και να μυρίζει σαν καπνός και να έχει γεύση καπνού. Ε, αυτό ιδιαίτερα για να μην είναι ελκυστικός προς τους νέους. μεταξύ του 2005 και 2011 με τις απαγορεύσεις του δημόσιου καπνίσματος είδαμε μείωση από το 39% στο 33% ε, του ποσοστού των νέων που καπνίζουν. Και πάλι βέβαια είναι ψηλό, μπορεί να βελτιωθεί και χρειάζονται περισσότερα μέτρα επιγόντως. Να συγχαρώ την Ιρλανδική Προεδρία γιατί ήταν εντυπωσιακό που ε, προάσπισαν ε, υποστήριξαν μάλλον τέτοιου είδου προτάσει τον περασμένο μήνα Συμβούλιο. Είπα η Ιρλανδία ότι αν το καπνό ήταν καινούριο προϊόν δεν θα έμπαινε ποτέ στην αγορά, δεν θα είχαν εμπορίε ποτέ. Ε, Ευχαριστώ. Η συνάδελφος ήδη αναφέρθηκε στο βασικό μας στόχο, δηλαδή καλύτερη υγεία των Ευρωπαίων ε, πολιτών. Λέει κυρία Χούμπνερ, υπάρχουν στοιχεία που εκλείπουν, που λείπουν ακόμα. Θα πρέπει να υπάρξει η σωστή κατάρτιση και εκπαίδευση προς αυτή την κατεύθυνση. Μιλάμε για την αρχή της επικουρικότητας, αλλά στα διάφορα κράτη-μέλη έχουμε και διαφορετικά όρια ηλικίας ως προς τη διαθεσιμότητα του καπνού. Ίσως θα πρέπει να μιλάμε για τα 18 χρόνια, για όριο 18 ετών παντού. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν καπνιστές οι οποίοι ασθενούν αργότερα. Γιατί δεν υπάρχει ένα διαφορετικό σύστημα ασφάλισης για τους καπνιστές. Ως προς την τηλεπόληση είναι πολύ εύκολη. Αν κάποιος είναι, και, είναι 14, μπορεί να βάλει στο κατάλληλο τετραγωνίδιο, στο σχετικό τετραγωνίδιο, την είναι 21, ποιος θα το ελέγξει αυτό. Εάν θέλουμε λοιπόν να καταπολεμήσουμε τη χρήση καπνού και οι νέοι μας είναι υγιείς, θα πρέπει να καταπολεμήσουμε και την τηλεπόληση. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν δελαστικά ε, πακέτα που μοιάζουν με κραγιόν, με γλύκισμα ή με οτιδήποτε άλλο. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριος Παρνιό, έχουμε ε, δυστυχώς ξεπεράσει τα εμπορικά όρια σε έναν πολιτισμένο κόσμο. Πρόκειται για μία βιομηχανία του εγκλήματος, διότι ο εθισμός των καπνό δημιουργεί 6 εκατομμύρια θύματα στον κόσμο, 800.000 στην Ευρώπη και θα φτάσει τα 8 εκατομμύρια. Για να αντιστρέψουμε αυτή την ολέθρια τάση θα πρέπει να προβάλλουμε συγκεκριμένα μέτρα εμείς ως πολιτικό και να προβούμε και στην αυτοκριτική μας. Ας μην είμαστε υποκριτές. Μιλάμε για την προάσπιση των ε, λιανοπολιτών ή των καλλιεργητών. Ας σταματήσουμε με αυτή μας τη στάση που είναι καθαρά πελατιοκρατική στάση. Θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτή την πολύ καλή οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και που υποστήριξε και η συγγήτριά μας. Θα ήθελα να υποβάλω μερικές τροπολογίες για να ενισχύσω το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας σε όλα τα προϊόντα καπνού και αυτό αφορά και τα αρώματα εθισμού, τη σήμανση καθώς και το μέγεθος. Και ας μην επιτρέπουμε περαιτέρω παράγωγα προϊόντα όπως αυτά τα τσιγάρα slim, τα οποία είναι δελεαστικά. Κα, Πρόεδρε, ευχαριστώ. κύριε και κύριοι, συμφωνώ με τα περισσότερα από όσα λέχθηκαν για τις αρνητικές συνέπειες του καπνού. Είμαι γιατρός και καταλαβαίνω πολύ καλά αυτά που λέτε. Και συμφωνώ με τα μέτρα προστασίας ανηλίκων και παιδιών από όλα τα ναρκωτικά επίσης, όχι μόνο τον καπνό. Η πολιτική της Ένωσης δεν θα πρέπει να λαμβάνονται, να, η πολιτική συνένωση δεν πρέπει να ασκείται μόνο στη βάση αποφάσεων που προέρχονται από τις Βρυξέλλες. Πολλοί συμφωνούν μαζί μου. Η κυβέρνηση της τσεχικής δημοκρατίας, το κοινοβούλιο, έχουν επίσης λάβει αποφάσεις. Η συγγήτρια, καθώς και άλλοι συνάδελφοι, είπαν καθαρά ότι οι χώρες μέλη είναι ικανές να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για να προστατεύσουν τους πολίτες τους από τις αρνητικές συνέπειε του καπνού. Είναι πολιτικός ο λόγος μόνο εναρμόνισης δηλαδή της προστασίας αυτής από τις Βρυξέλλες. Οι χώρες μέλη και τα κοινοβούλια τους δεν είναι λιγότερο ευφύ ή υπεύθυνα από ότι είμαστε εμείς εδώ στις Βρυξέλλες. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και θα ήθελα να πω ότι ήταν πολύ θαραλέα και χρειαζόμαστε πολύ φάρος διότι τα λόμπι όχι μόνο επισκέπτονται το Κοινοβουλίο, αλλά μας ε, ε, κατακλείζουν με επιστολές και πολλοί ε, αναφέρουν τη δυσκολία με την αρχή της επικουρικότητας. Ακούσατε τι είπε και ο προλαλής σας. Είναι κάτι το ολέθριο. Κάθε χρόνο πεθαίνουν 700.000 καταναλωτές και γι' αυτό η καπνοβιομηχανία χρειάζεται κάθε χρόνο νέους καταναλωτές. Υπάρχουν ειδικέ γεύσεις που καθιστούν το κάπνισμα ευκολότερο, πιο δελεαστικό. Υπάρχουν πολλά, ε, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο δέλεαρ της αγοράς και γι' αυτό θα πρέπει να προωθήσουμε την πρόταση της Επιτροπής η Επιτροπή μας ε, θα πρέπει να ε, δώσει μεγάλη μάχη υπέρ των ε, Ευρωπαίων πολιτών στο τομέα της υγείας. Πιλάρα Γιώσο. Ό,τι είναι υπέρ της υγείας πρέπει να το υποστηρίζουμε πάντοτε. Νομίζω ότι υπόθηκε ότι ήταν υποθεί, αλλά να υπογραμμίσω κάτι που είπα και όταν ήταν εδώ ο Επιτροπός. Η οδηγία θα πρέπει να εναρμονιστεί με το πρωτόκολλο για την κατάρριση του λαθρεμπορίου ε, προέντων καπνού. Και το άρθρο 14 της οδηγίας ε, δεν είναι ευθυγραμμισμένο με το πρωτόκολλο. Το πρωτόκολλο υιοθετήθηκε τον Νοέμβριο του 2012, ψηφίστηκε υπέρ από τα 26 από τα 27 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με άλλες 140 χώρες του κόσμου. Θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν τα κείμενα της οδηγίας με το του πρωτοκόλου. Θα πρέπει ο κώδικας να είναι ενιαίος, ασφαλής, σίγουρος ε, ε και να αφορά όλα τα προϊόντα καπνού. Ε, επίσης, είναι πολύ σημαντική η εκπαίδευση και οι, οι ενημερωτικές εκστρατείες του κοινού. Είναι πολύ σημαντικό να εκπαιδεύουμε τα παιδιά στα σχολεία και, και τον ευρύτερο πληθυσμό. Σε ό,τι αφορά τα όσα είπε ο κ. Λίσε, ε, η επιδοτήσεις είναι επιδοτήσεις σε μια καλλιέργεια, όχι στον καπνό τον ίδιο. Είναι ε, όπως επιδοτήσεις για τα, το ζαχαρότευλα που και ασφαλώς παράγουν και ζάχαρη που κάνει και αυτή κακό. Ευχαριστώ. Σοφία Κονή. Θα ήθελα λίγο περισσότερο χρόνο, Πρόεδρε, γιατί μιλώ εξ ονόματος της ε, κυρίας Γκροστέτ και μετά θα προσθέσω ε, ορισμένες σκέψεις δικές μου. 1,5 λεπτό, λέει ο πρόεδρος. Θα προσπαθήσω, θα προσπαθήσω. Η μελλοντική οδηγία θα πρέπει να δει τη ρίζα της κακοδαιμονίας που υπενθύμησαν πάρα πολύ και η Φρανσουάζ Γκροστέτ που δεν είναι εδώ γιατί χρειάστηκε να φύγει για μια άλλη συνεδρίαση θα ήθελε να τα δούμε τα θέματα πολλαπλώς. Πρόληψη, οι εκστρατείες πρόληψης δεν επαρκούν. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει μία ε, ευαισθητοποίηση η οποία να είναι στοχοθετημένη. Πέρα από αυτά που έχουν γίνει μέχρι τούδε για να επιλέξουμε μέσα διάδοσης που να έχουν σαν βασικό στόχο τους νέους οι, μαζικέ οι μαζικές εκστρατείες ε, μπορούν να έχουν πολύ καλή σχέση κόστους ωφελίας σε σχέση με άλλες παρεμβατικές δράσεις στον ε, τομέα της υγείας και καταπολέμησης της χρήσης καπνού. Θα πρέπει... Θα ήθελα να προσθέσω και την κατάρτιση στα σχόλια. Θα πρέπει να επιβάλλουμε στα κράτη-μέλη να προωθήσουν αυτή την εκστρατεία κατά του καπνού στα σχολεία. Να εξηγούμε στα παιδιά πόσο επικίνδυνη είναι η χρήση. Ως προς τα ηλεκτρονικά τσιγάρα θα πρέπει η Επιτροπή να μας πει κατά πόσο διαθέτει επιστημονικές μελέτες για να πλαισιώσουμε καλύτερα αυτό το προϊόν. Γιατί σε ορισμένα κράτη θεωρούνται απλώς τσιγάρα, ενώ σε άλλα φαρμακευτικός σκεύασμα μεταξύ άλλων. Χρειαζόμαστε περαιτέρω στοιχεία, σήμανση. Δεν θα αλλάξουν τα πράγματα αν βάλουμε εικόνες. Σήμερα η καπνοβιομηχανία πολύ υπέροχες θήκες, πανέμορφες, έτσι ώστε να ε, κρύψουμε αυτές τις εικόνες και τη σήμανση. Άρα θα πρέπει να, αυξήσουμε τιμή ε, καπνού. Μα μένουν 10 λεπτά και θέλουμε να απαντήσει και η Κομισιόν, καθώ επίση να λάβει το λόγο η εισηγήτρια. Να μπορέσει δηλαδή να απαντήσει ενδεχομένω. Η συζήτηση ήταν χρήσιμη. Για τα ηλεκτρονικά σιγαρέτα είναι πιο πολύ προϊόντα ατμοποίησης ή εξάτμισης το, της νοικοτήνης. Δεν ξέρω τέλος πάντων εάν όντως το προϊόν ο, υπάγεται σε τούτην εδώ την οδηγία. Αυτά τα ηλεκτρονικά σιγαρέτα δηλαδή. Έμαθα τελευταία ότι πολλοί πρώην καπνιστές τα χρησιμοποιούν για να ξεσυνηθίσουν το κάπνισμα και ότι δεν αρχίζουν την επαφή με το κάπνισμα οι νεαροί καπνιστές. Βέβαια, αντιλαμβάνομαι ότι ενδέχεται η καπνοβιομηχανία ενδιαφέρεται να αποσυρθεί το προϊόν αυτό το δυνατόν συντομότερο από την αγορά. Πάντως, όπως ακούσα, θα ανατεθεί μελέτη και νομίζω ότι κάτι τέτοιο ενδιαφέρει πολλούς. Πρόκειται βέβαια για σκληρά εμπορικά συμφέροντα που θέλουν να φύγει από την αγορά το προϊόν αυτό, το ηλεκτρονικό σιγαρέτο. Πάντως επαναλαμβάνω ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη σήμερα η συζήτηση και μια και έχουμε φτάσει εδώ θα δώσω το λόγο στον κύριο Ντόμινικ Στίχελ. Πέντε λεπτά είναι δυνατόν, ξέρω ότι είναι, σας ζητώ το αδύνατον, αλλά έτσι θέλω να μπορέσει και η εισηγήτρια να απαντήσει. Γιατί οι κυβερνήσεις μπορούν να προχωρήσουν περισσότερο στο plain packaging. Ναι, στην αιτιολογική σκέψη 41 το λέμε καθαρά και στην παράγραφο 24.3 θα είναι δυνατό. Γιατί ρυθμίζουμε το SNUS. Με εξαίρεση μόνο της Σουηδικής κυβέρνησης αναφέρεται στην διάθεση στην αγορά και όχι σε ρύθμιση του ίδιου του προϊόντος. Γι' αυτό ρυθμίζουμε την επισήμανση και επεκτείνουμε την ίδια ε, ρύθμιση και σε αυτό. Διαμεθοριακές πωλήσει, από, τηλεπολίσεις δηλαδή, έχετε τη σχετική ρύθμιση. Νομίζουμε πάντως ότι η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να αποτελέσει το λιγότερο αποτελεσματικό μέσον για τον έλεγχο αυτών των τηλεπολίσεων και ενδέχεται μάλιστα η πρότασή μας να είναι πιο συμβατή έτσι με την ε, ισχύουσα νομοθεσία. Ε, ηλεκτρονικά σιγάρετα που έφτιαξαν πολλοί συναδελφοί σα γιατί μπαίνει στην οδηγία προϊόντων καπνού. Η νοικοτήνη στα ηλεκτρονικά σιγαρέτα προέρχεται από τα τσιγάρα. Είναι υποκατάστατο προϊόν για τον καπνό. Θεωρούμε λοιπόν ότι υπάγεται στην οδηγία. Υπάρχουν Πολλέ βέβαια ανησυχίε γύρω από την ασφάλεια και γι' αυτό χρειάζεται να δραστηριοποιηθούμε. Μιλήσαν ορισμένοι και για το κίνδυνο ε, θανάτων παιδιών εάν ε, πιούν το περιεχόμενο του κυλίνδρου αυτού. Βέβαια αρχικά Αρχικά τα ηλεκτρονικά σιγαρέτα τα χρησιμοποίησαν καπνιστές ενήλικοι για να ε, ξεσυνηθίσουν το κάπνισμα, ωστόσο διαπίστωσε ας πούμε ουγγρική μελέτη ε, ε, του 2012 ο 13-15% των νεαρών καπνιστών χρησιμοποίησαν τα ηλεκτρονικά σιγαρέτα για να ξεκινήσουν. Αρχίζουν λοιπόν και εθίζονται και μετά περνούν από τα ηλεκτρονικά σιγαρέτα στα κανονικά. Παρόμοια μελέτη στην Πολωνία έδειξε ότι 20% των Πολωνών νέων έχουν πειραματιστεί με ηλεκτρονικά σιγαρέτα. Τελευταίο θέμα. Δεν θέλουμε να δούμε τα ηλεκτρονικά σιγαρέτα να αποχωρούν από την αγορά. Αντιθέτως, εάν πρόκειται για αποτελεσματικό μέσο που θα βοηθήσει τους καπνιστές να ε, απομακρυνθούν από το να ξεσυνηθίσουν το κάπνισμα, να το υποστηρίξουμε. Όμως θεωρούμε ότι πρέπει να είναι ρυθμισμένο και να λειτουργεί μέσα σε ε, ελεγχόμενο περιβάλλον, δηλαδή στα φαρμακεία, το οποίο θα εξασφαλίσει και την, ε, τον ισότιμο ανταγωνισμό με άλλα μέσα ε, υποκατάστασης της νοικοτήνης. Είναι ζήτημα λοιπόν χορήγησης του προϊόντος. Η μόνη διαφορά μεταξύ ηλεκτρονικών ε, σιγαρέτων, σπρέι ή ε, αυτού αυτό που βάζουμε πάνω στην επιδερμίδα δηλαδή, για τη διοχέτευση της νοικοτήνης είναι αυτό. Τώρα, για τα άλλα, 50% της αύξησης των ε, slim, των σιγαρέτων slim, των λεπτών αυτών σιγαρέτων, 50% αύξηση τα τελευταία χρόνια, τέτοια προϊόντα που μοιάζουν σαν να είναι το κραγιόν των χιλιών. Αυτά όλα έχουν ε, έτσι ένα χαρακτήρα chic, κομψό κτλ. Και, και αυτό είναι ιδιαίτερα ελκυστικά για τους νέους και τις νέες τα ε, πουράκια τώρα. Μπορεί όντω μέσω αυτών να υπάρξει ένας τρόπος καταστατήγησης της νομοθεσίας. Νομίζουμε όμως ότι μπορούμε να αντιδράσουμε εάν δούμε ότι αυξάνεται η κατανάλωση ε, πουρακίων, να πούμε έτσι, τότε μπορούμε να ε, αντιδράσουμε. Απαγόρευση του display. Αυτό μπορεί να είναι δυνατόν. Ωστόσο, μπαίνει στην οδηγία προϊόντων και όχι οδηγία περί Άρα δεν εντάσσεται εδώ. Νομίζουμε ότι πρέπει να μπει στην οδηγία για τις διαφημίσεις. Αν μπορούμε τώρα να ρυθμίσουμε περισσότερο τις διαφημίσεις, για τους ίδιους λόγους που είπα, πρόκειται για οδηγία αυτή που σας προτείνουμε εδώ δηλαδή, η οποία ρυθμίζεται από των προϊόντων και όχι τις διαφημίσεις τους. Επίσης, ακούστηκε μια ερώτηση για composite cans, για κουτιά ε, σαν κονσέρβες ας πούμε. Γιατί δεν προτείνουμε ε, τα, το, το, το καπνό για τσιγάρα μέσα σε φακελάκια. Έχουμε μόνο περιλάβει τον καπνό πίπας. Υπάρχουν διαφορές εδώ και διαφορετικά, διαφορετικές συσκευασίες, διαφορετικά δοχεία, είτε σε φακέλους είτε σε ε, κονσέρβες. Επίσης, όταν βγείτε έξω, δεν θα πάρετε στην τσέπη σας 200 γραμμάρια, ε, κουτί δηλαδή 200 γραμμαρίων καπνού στη τσέπη, δεν νομίζω. Τέλος, περιορισμοί ηλικίας, αν μπορούμε να το βάλουμε με τη νομική βάση του άρθρου 14. Νομίζουμε ότι αυτό δεν είναι δυνατόν και είναι αρμοδιότητα των χωρών μελών. Επομένως δεν θα πρέπει να δράσουμε στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Μιλήσατε και για τα υγρά όταν καταποθούν αλλά και τι γίνεται με όλες αυτές τις γόπες που ε, βρίσκει κανείς στους παιδικούς, ε, στις ε, παιδικές χαρές κλπ. Φανταστείτε, θα έπρεπε λοιπόν αν είναι να τα απαγορεύσουμε, θα έπρεπε να απαγορεύσουμε κάθε κατανάλωση σιγαρέτων. Λαμβάνει το λόγο τώρα η συγκίτρια. Θα είμαι σύντομη. Ευχαριστώ τους και τις συναδέλφους για τα σχόλιά τους. Οι περισσότεροι στηρίζουν την νομοθεσία, υπάρχουν κάποια κρεμή θέματα. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, για παράδειγμα, χρειάζεται να συζητηθούν περισσότερο. Πρέπει να ακούσουμε τους εμπειρογνώμονες, γιατί ε, θέλουμε να εγκρίνουμε την πιο κατάλληλη νομοθεσία για αυτά. Ίσως θα οργανώσω ένα εργαστήρι, μια ακρόαση, για αυτό ακριβώ το θέμα, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Για τις πωλήσει μέσω ίντερνετ, η κυρία Χίμπνερ είπε πω είναι προβληματικές σε ορισμένες χώρες Γερμανία παράδειγμα, μπορεί κανείς να πάρει και δωρεάν τσιγάρα από το ίντερνετ να αποκτήσει. Σε άλλες χώρες όπως την Ελλάδα ε, τσιγάρα μοιράζονται δωρεάν σε δισκοτέ και nightclubs ε, στους νέους. Πρέπει να τα δούμε αυτά τα θέματα. Σε ό,τι αφορά τα μεντόλ, τα τσιγάρα με, μέντα, με μεντόλ. Γιατί στον Καναδά και τις ΗΠΑ δεν έχουν απαγορευτεί. Δεν ξέρω για τον Καναδά. Έχω μιλήσει όμως με ανθρώπους της ΗΠΑ. Στις Πολιτεία ειλικρινά, γιατί η FDA ε, δεν τα απαγόρευσε εξαιτία πιέσεων που δέχθηκε, όχι για επιστημονικούς λόγους. Η Επιστημονική Επιτροπή στι ΗΠΑ ε, ε, είχε προτείνει ε, ε να απαγορευτούν. γιατί, γιατί ε, το, το μεντόλ κάνει πιο ελκυστικά τα τσιγάρα και ε, αυξάνει και την εισπνοή τους, τη δυνατότητα εισπνοής. Ε, δεν συμπερέλαβαν όμως τα τσιγάρα μεντόλ ε, στις ΗΠΑ στην απαγόρευση για τα, τις ουσίες, όμως ε, κάποιοι έχουν προσφύγει εναντίον τη Κυβέρνησης των ΗΠΑ στο δικαστήριο για λόγους ανταγωνισμού, διότι είναι σαν να υπάρχει μια διακριτική μεταχείριση εναντίον αυτής τη ουσία. Ε, ας είμαστε προσεκτικοί, με την εξαίρεση μιας ουσίας μπορεί να καταπέσει όλη η νομοθεσία μας. Ας είμαστε πολύ προσεκτικοί να μην επιτρέψουμε στα διάφορα λόμπι από την πίσω πόρτα να ε, πλήξουν το υπόλοιπο έργο μας. Τέλος. Όχι, νομίζω πως τα κάλυψε όλα. Α, για τις εξτρα, πληροφορικές εκστρατείες. Ναι, ασφαλώς και χρειαζόμαστε. Αλλά κυρία Οκόνη, δεν έχουμε την εξουσία να υπαγορεύσουμε στις κυβερνήσεις ε, να κάνουν το α ή το β με το εκπαιδευτικό του σύστημα. Ε, εμείς είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εδώ. Ασφαλώς, οι εικόνες, ε, οι εικόνες πάνω στα πακέτα ε, δεν θα αποτρέψουν όλους τους νέους από το να καπνίζουν. Αλλά οι εμπειρογνώμονες, οι γιατροί, ειδικοί λένε ότι τέτοιου είδους εικόνες έχουν επιπτώσεις έχουν αποτέλεσμα σε ορισμένους νέους. Και ορισμένους νέους σημαίνει ορισμένες ζωές. Ε, η Κομισιόν μας έχει πει ότι το 94% των καπνιστών ξεκινάνε πριν τα 25 χρόνια τους. Συνεπώς είναι πολύ σημαντικό να εστιάσουμε στους νέους για να μην γίνουν καπνιστές. Εγώ δεν καπνίζω ε, παρόλο που κουβαλάω ένα κάρο πακέτα μαζί μου. Ε, δεν ξεκίνησα να καπνίζω. Ε, ας ε, επιλέξουμε να έχουμε ένα συνολικό σύστημα, αλλά χωρίς να λέμε μην κάνουμε αυτό γιατί θα πρέπει να κάνουμε και το άλλο και δεν μπορούμε να κάνουμε το άλλο κλπ. Ας ε, μην ακούμε τα λόμπι, χρειαζόμαστε ένα, μια πλήρη νομοθεσία για τα προϊόντα καπνού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πραγματικά ενδιαφέροντα λόγια. Θα ξαναβρεθούμε στις 3. Εδώ λίγη συζήτηση του θέματος αυτού και